Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία για σήμερα. Έκθεση για το Αφγανιστάν του κυρίου Αρλάκη. Σας παρακαλώ. Να. Ετοιμάσετε τις κάρτες σας στο μηχάνημα. Ο κύριος Μάντνερ για το κανονισμό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω με κάποια πράγματα σχετικά με τις ψηφοφορίες. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες να κάνουμε. Πριν από μισή ώρα πήραμε 400 τροπολογίες και πριν από δύο ώρες πιο μπροστά άλλο ένα πλήθος 300 τροπολογιών. Δεν νομίζω ότι έχουμε ε, προετοιμαστεί για όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει τουλάχιστον 24 ώρες πιο πριν να ε, έχουμε τις τροπολογίες στη διάθεσή μας. Και θα ήθελα πραγματικά να το λάβουμε υπόψη αυτό, τη δική μας προετοιμασία, αλλά και τη, τους βοηθούς ε, και τους συνεργάτες μας που δουλεύουν ε, λοιπόν πρέπει και αυτοί να προετοιμάσουν τα πράγματα. Πράσι. Λοιπόν, η λίστα είναι έτοιμη, στο τε... θα είναι έτοιμη εν πάση περιπτώσει, λυπούμε πάρα πολύ, σε αυτό το δυσάρεστο επεισόδιο. Θα κοιτάξουμε να το αποφύγουμε ξανά. Λοιπόν, ε, ξεκινάμε την ψηφοφορία, αν έχετε την κάρτα σας. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Δεν είμαι σίγουρος για το τι έχω διαπιστώσει με τα μάτια μου. Λοιπόν, ελέγχουμε την 103. 57, 58 ψήφισαν. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές. Ε, μου φαίνεται να εγκρίνεται. Λοιπόν, έλεγχος για την 106 αρχίζει ψηφοφορία. 56 ψηφίσαντες. Απορρίπτεται. 32-24. 107 έχει αποσυρθεί, 108 δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Δεν συμφωνείτε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 108 και αρχίζει η ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Πέρας ψηφοφορίας. ψηφοφορίας. 34-27. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος. 122. Αρχίζει η ψηφοφορία. 122. «32 όχι, 27 ναι, απορρίπτεται, 123 υπέρ». «Κατά» αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 αποσύρθηκε. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές θα, θα έλεγα ότι απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 127. 62 ψηφίσαντες. Απορρίπτεται. 33 κατά και 28 υπέρ. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 πίπτη, 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται να έχει απορριφθεί απορρίφθηκε ωραία 133 υπέρ Α, ναι, ναι, ναι, απορρίψαμε την 131, πάμε στην 132, υπέρ. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133. Α, όχι. Εγκρίθηκε 131. 134 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε unblock τις τροπολογίες 135, 136, 137, 138, 139, 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκαν. Έλεγχο. Ωραία. Ξεκινάει ο έλεγχος για τις τροπολογίες σαν μπλοκ από τις 135, την 135 στην 140 και αρχίζει η ψηφοφορία. 64, 64 schede, 62 voti espressi. 62 ψηφίσαντες πέρα της, ψηφοφο... Ε, πέρα της ψηφοφορίας. Περνάει 38-24. 141. Δεν ψηφίζουμε. 142 ε, αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε ευτυχώς unblock 143 ως 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν εξήντα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, να ελέγξουμε την 164 γιατί και εγώ έχω αμφιβολία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 164. 63 ψηφίσαντες. Εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται η 166. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αποσύρθηκε 168. Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά. Δεν είδα καλά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 173, αρχίζει η ψηφοφορία. Παρακαλώ να σηκώνετε το, τα χέρια σας καλά, γιατί χάνουμε ώρα με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. 66 ε, κάρτες ε. Ε, ε, Λοιπόν, 6. 52-7 λοιπόν. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. εγώ λέω όχι. Αλλά λίγα χέρια σηκωθήκανε. Λοιπόν, τρέφω εμπιστοσύνη στις μαντικές μου ικανότητες. Παρακαλώ, σηκώντε τα χέρια σας. 188 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εδώ ήταν καθαρά τα πράγματα εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές αμφιβολία αμφιβολία ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 190 190. 62 ψηφίσαντες. 63. 34-29 εγκρίνεται. 192 υπέρ κατά αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 194 υπέρ κατά αποχές θα λέγω ότι εγκρίνεται όχι Λοιπόν, δεύτερο τμήμα της 194. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 48 όχι, 18 ναι. 195 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ. Όχι, όχι. Πέρασε 199. Ωραία, λέει ο πρόεδρος, διορθώνομαι. Η 200 έχει καταπέσει. Πάμε στη 202. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εγώ το βλέπω να εγκρίνεται. Άμα δεν σηκώνω τα χέρια τι να κάνω, Λέω ο πρόεδρος. 204 λοιπόν. 203, 203 διορθώνει το πρόεδρος. Ε, ναι, αλλά και οι δύο διαγραφές είναι. Α, είναι το ίδιο κείμενο, ωραία. Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μου το έχετε γράψει. 204 λοιπόν. Καταπίπτουν οι 204 και 205. Λοιπόν, 208 σε δύο τμήματα. 208 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρόεδρε. Για την 202 μπορώ να ζητήσω να ξαναψηφίσουμε. Εγώ το, το να το ψηφίσουμε, αλλά μου είπανε τη γραμματεία ότι είναι το ίδιο πράγμα, 202-203. Ήδη ψηφίστηκε λοιπόν. 208, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται να έχει εγκριθεί. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 220 σας παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 35 υπέρ 27 κατά. 221 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ. Α, είναι το ίδιο. Ε, μα δεν μου το γράφετε ότι είναι το ίδιο πράγμα. 226 υπέρ. Α, τότε να πάμε στην 228 λέει ο πρόεδρος. 228 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 αποχές απορρίπτεται 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 245, 246 tutti, eh, 246. 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 259 υπέρ Διακόπτουμε την 259 γιατί θέλει το λόγο ο κύριος Δαβίντ. Πρόεδρε, εδώ βλέπω ότι η 255 πρέπει να ψηφιστεί εάν απορριφθεί η προηγούμενη. Αλλά την εγκρίναμε την προηγούμενη. Συνεπώς δεν πρέπει να ψηφίζουμε επί της 255. Ma è stata adottata?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 αποχές εγκρίνεται 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 262 αποσύρθηκε 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές μα εγώ το βλέπω να απορρίπτεται άρα δεν σηκώνετε τα χέρια σας λοιπόν 265 να ελέγξουμε εντάξει αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία για τη 265 Πέρας ψηφοφορία. 33 ναι, 32 όχι, εγκρίνεται. Λοιπόν, συμβιβασμός 12 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 13 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 280 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 14 τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα έλεγα. Να το ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα του συμβιβασμού 14 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 34 υπέρ 28 κατά εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.91 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το ίδιο και 293 που δεν θα την ψηφίσουμε. 294 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 296 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 301 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 15, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 307, υπέρ. η προφορική τροπολογία είναι 306, εντάξει. Προφορική τροπολογία για την 306, υπέρ. Κατά. Ε, ο πρόεδρος, να ελέγξουμε, δεν είδα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 306 πρόκειται για προφορική τροπολογία. 66 schede, 63 votanti, chiusa la 26 όχι 33, ναι πέρασε λοιπόν. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 309 υπέρ. Κατά. Αποχές μου φαίνεται να εγκρίθηκε. Δεν είμαι όμως πανσίγουρος. Έναξε, ωραία. 310 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 313 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 312 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 320 υπέρ κατά αποχές α δεν ξέρω ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία για την 320 ε, σήμερα δεν έχετε καμία όρεξη να σηκώνετε το χέρι σας, λέει ο πρόεδρος. 320. Πέρα στις ψηφοφορίες. 28, όχι 36, ναι εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 16, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 327, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 320 Α, 330, 330 λέει ο πρόεδρος, υπέρ κατά αποχές. Μπα, θα έλεγα ότι απορρίφθηκε. Όχι, τι λέτε. Να το ελέγξουμε λοιπόν. 330. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 330. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 332 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 333 θέλετε να ελέγξουμε την 332 εντάξει ήταν σαφές λοιπόν πάμε στην 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 335 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 334 Allora, dobbiamo chiedere all'onorevole Scholz se è d'accordo con la proposta del relatore riguardo alle... Συμφωνεί ο κύριος Σόλτς με την πρόταση του εισηγητή για την 334. Κύριε Σόλτς, συμφωνείτε? Ωραία, να ψηφίσουμε έτσι πως το λέμε λοιπόν. 334, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Α, ε, τι να κάνω, μονάζιγα πρέπει να το παίζω. 336 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 337 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 338 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 342 και 343 είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 344 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 18, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 353 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 354 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 355 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εδώ έχουμε, α δεν ψηφίζουμε 358 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 359 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 361 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα... Έχουμε λοιπόν ένα αίτημα να ψηφίσουμε το αυθεντικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ο Αρλάκη. Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Δεν ήταν καθόλου σαφές. Ε, τι να πω, ήδη ψηφίσαμε. Μα είχαν σηκωθεί λίγα χέρια. Ε, το ξέρω, αυτό λέω συνέχεια, λέω ο πρόεδρος. Γι' αυτό λέω και εγώ, λέει ο κύριος Αρλάκη, ότι δεν ήταν καθαρά. δεν ήθιστε γιατί τελειώσαμε την ψηφοφορία για, την τροπολογία στα τρία τμήματα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ας κάνουμε μία εξαίρεση. Αλλά δεν θέλω να επαναληφθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει, έχουμε ψηφίσει και... Λοιπόν, να ξαναψηφίσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας για την παράγραφο 57. Αρχίζει η ψηφοφορία. Για το δεύτερο τμήμα. Πέρα στις ψηφοφορίες. 48, όχι 17, ναι. Λοιπόν, 364 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 367 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα έλεγα 368 υπέρ Α, 367 αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. 47-18 λοιπόν 369 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ είναι προφορική τροπολογία κατά αποχές εγκρίνεται 371. Η 70 εγκρίθηκε. Α, στη 373 λοιπόν πάμε. Υπέρ της 373. Υπέρ της 373. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 377 <coughs> υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίφθηκε 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 380 υπέρ κατά αποχές. Μπα, τι να πω λέει ο πρόεδρος και εγώ λέω ότι απορρίφθηκε. 381 υπέρ. Υπέρ της 381 κατά αποχές. Εγκρίνεται. 382 και 383 είναι ίδιες υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 384 υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν την ψηφίζουμε γιατί εγκρίναμε την προηγούμενη. 386 λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 387 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 388 υπέρ. Κατά αποχές. Μου φαίνεται να έχει απορριφθεί. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Ωραία. 388 την ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 389 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δέκα υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται να εγκρίσκει.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 αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 29 αρχίζει ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της 29 πέρας ψηφοφορίας. 33 κατά απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές μα λέει ο πρόεδρος εγώ λέω ότι απορρίφθηκε αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος συμβιβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέχρι και τις 47 είναι όλες ίδιες. Λοιπόν 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίφθηκε 50 υπέρ κατά αμφιβολία, αμφιβολία για την 50 ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 50 ηλεκτρονικά για την 50 Chiusa la votazione. Πέρας ψηφοφορίας. 47-19. <laughs> Εγκρίνεται. 47-19. 51 υπέρ. Κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Αποσύρθηκε 52-53 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 25 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με αμφιβολίες 59 Ωραία, να μην λέω τι αμφιβολίες μου. Καλά, εντάξει. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 58. Πέρας ψηφοφορίας. 44 όχι, 14 ναι. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 26 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 Α, ζητήσατε έλεγχο για την 67. Ωραία, να ελέγξουμε την 67 και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μπλοκ. Από το 1 ως το 12 εκτός από την 9. Είπαμε 1 ως 12 εκτός της 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικά, πρόεδρε ο Αρλάκη. Ονομαστική ψηφοφορία ζητώ, λέει ο κύριος Αρλάκη. Μπορούμε να τη δεχτούμε λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Για την έκθεση Αρλάκη. Δύο δεν ψήφισαν. Ένας δεν ψήφισε. Πέρα της ψηφοφορίας. 60 υπέρ, ένας κατά, πέντε αποχές. Ευχαριστώ τον εισηγητή, συγχαρητήρια, μεγάλη πλειοψηφία. Ο κύριο Βανόρντεν. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση επί της διαδικασίας. Μόλις ε, ψηφίσαμε μια έκθεση με 400 περίπου τροπολογίες και η επόμενη έκθεση άλλες τόσες θα έχει περίπου. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος δουλειάς αυτός. Όταν υπάρχουν τόσο πολλές τροπολογίες, κάτι άλλο θα πρέπει να κάνουμε. Ίσως θα πρέπει όταν υπάρχουν τόσο πολλές τροπολογίες ο εισηγητής ενδεχομένως να αναθεωρήσει, να ανασυνθέσει να ξαναφτιάξει την έκθεσή του για να προτείνει κάτι καινούριο ε, ε, ε, αλλά το να ψηφίζουμε 400 και τροπολογίες είναι λίγο περίεργος τρόπος να διεκπαιρεώνουμε τα... τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Βίγενιν και μετανέιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως όταν έχουμε τέτοιου είδους εκθέσεις με τόσες τροπολογίες δεν είναι εύκολα τα πράγματα αλλά μιλάμε για διετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μιλάμε για σοβαρά θέματα ο εισηγητής και οι σκιώδες ε, καταβάλαν μεγάλες προσπάθειες για να προετοιμάσουν τέλο πάντων μια ψηφοφορία για να αναζητήσουν συμβαστικές λύσεις και Και εγώ λέω ότι θα πρέπει και την έκθεση αυτή να την ψηφίσουμε τον ίδιο τρόπο που κάναμε πριν, παρόλο που μπορεί να κουραστήκαμε από την έκθεση για το Αφγανιστάν. Σήμερα λοιπόν θα ψηφίσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, θέλουμε η έκθεση αυτή να πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αν αναβάλουμε σήμερα δεν την ψηφοφορία δεν θα μπορέσουμε έγκαιρα να την τελειώσουμε ώστε να πάει στο, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Η κυρία Νέιτς, πρόεδρε, συνάδελφοι, ε, πραγματικά έχω αντίστοιχε ανησυχίε με αυτέ του συναδέλφου Βαν Όρντεν όταν ε, για το τεράστιο αριθμό τροπολογιών για τι εκθέσει αυτέ. Ε, δεν σχετίζεται αυτό βεβαίως με την ποιότητα ή την συνεκτικότητα των εκθέσεων αυτών καθεαυτών ε, ίσως ε, Κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να βελτιώσουν ακόμη και στις λεπτομέρειες το κείμενο και γι' αυτό ε, κάνουν τροπολογίες. Με αυτή την έννοια ίσως εμείς οι ίδιοι θα έπρεπε να αυτοπεριοριστούμε κατά κάποιο τρόπο και να μην καταθέτουμε τροπολογίες εάν δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να λογοκρίνω κανένα. Ο καθένας από μόνος το αποφασίζει. Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει δίκιο ο κύριος Βανόρντεν ότι είναι πάρα πολύ κουραστική όλη αυτή η ψηφοφορία λόγω του μεγάλου αριθμού των τροπολογιών. Αλλά είναι βέβαιο όμως κύριε Πρόεδρε ότι όλοι μας είχαμε τροπολογίες για αυτές τις εκθέσεις. Οι συνάδελφοι που είναι εδώ παρόντες κατέβαλαν μια τεράστια προσπάθεια. Θα έπρεπε λοιπόν να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία ούτω ώστε το θέμα να παραμείνει το Δεκέμβριο στην ολομέλεια και να λάβουμε στο μέλλον τα μέτρα για να μην είναι τόσο κουραστικά τα πράγματα. Σήμερα όμως πρέπει να ψηφίσουμε. Η ε, κυρία Χάπταλα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου που θα είναι ε, παρούσα η αρμοστία και τα λοιπά. Ιούνιο και Δεκέμβριο γίνεται κάτι τέτοιο. Θα ήταν ντροπή λοιπόν να μην πάει ε, το θέμα στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και οι, ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές. Λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε οπωσδήποτε σήμερα. Όλοι συμφωνούν μαζί σας κύριε Βανόρντε, πόσο μάλλον και ο πρόεδρος, ο οποίος πραγματικά κουράζεται πάρα πολύ όταν έχει 450 ψηφοφορίες και κάνει και λάθη πολλές φορές. Ο κανόνας όμως της δημοκρατίας επιβάλλει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις απόψεις. Σίγουρα ευκταίο θα ήταν, όπως ε, είπανε πολλοί και εγώ συμφωνώ μαζί τους, να βρούμε συμβιβαστικές φόρμουλες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 Η ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα της 47. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ναι, 18 όχι. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ και εγώ το περίμενα το περίμενα ηλεκτρονική για την 65 αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 65 πέρας ψηφοφορία 32, όχι, 28, ναι, απορρίφθηκε. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Είναι συμβατή με την 69. Υπέρ. Κατά. Εγώ λέω ότι εγκρίθηκε. Αλλά σηκώστε τα χέρια σας καλά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 και 76 είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγώ θα το έλεγχα αρχής ψηφοφορία για την 91 πέρας της ψηφοφορίες. 16-27 απορρίφθηκε. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 του εισηγητή. Πρώτο τμήμα. Α, όλο μαζί, με συγχωρείτε, όλο μαζί το ψηφίζουμε. Όλο, όλο μαζί λοιπόν, υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. 104 υπέρ. Κανένα δεν υπέρ της 104. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 118 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Η 115 έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 116 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 130 υπέρ κατά αποχές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 Έχω μία αμφιβολία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 135. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 28-26. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 11 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε το 150. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 55 όχι. Μα διάβασα τις σκέψεις σας, απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Μου κάνετε και αστιάκια βέβαια. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, μα θέλετε να με στρώσετε αγρίως στη δουλειά. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 155 ηλεκτρονικά. Μα έχω συναδέλφους οι οποίοι έχουν το, την κάρτα τους ε, στο μηχάνημα και δεν ψηφίζουν. Λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία. 27-27, δύσκολο, δύσκολο. Απορρίπτεται λοιπόν. 156 είναι ίδια με την 95, τις ψηφίζουμε και τις δύο. Η υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 40 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφ... Ε, ε, εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά Αποχές. Δεν το δω Η ηλεκτρονικά λοιπόν το, την 170. Πέρα της ψηφοφορίας. 49-10 εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 δύο τμήματα. 175 ωραία. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία της 175 που ζητούν οι σοσιαλιστές. 175 πέρα της ψηφοφορία. 34 ναι. Λοιπόν, πρόστιμο στους σοσιαλιστές γιατί με κάνανε να χάσω ώρα. Είχε περάσει. 176 σε δύο τμήματα. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Ο αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 14 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές ε, αυτό δεν το βλέπω. Ψηφίζουμε λοιπόν την 184 ηλεκτρονικά και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 15 Α, μάλιστα, απορρίφθηκε 185, ψηφίζουμε λοιπόν την 186, υπέρ της 186. Απορρίπτεται Συμβιβασμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 του εισηγητή συμβιβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 Σοσιαλιστική ομάδα ζητά ηλεκτρονικό έλεγχο, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 32 όχι. Δεύτερο πρόστιμο στη σοσιαλιστική ομάδα. 196 Για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, εδώ δεν είναι σαφές. Δεύτερο τμήμα της 197 λέει ο πρόεδρος. Chiusa la votazione. Ε... Πέρα στις ψηφοφορίες. Εμπερνά 28-28. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 207. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη 207. 207 πέρας της ψηφοφορίας 41 όχι 16 ναι 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 συγγνώμη συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τη 212. Πέρας ψηφοφορίας. 2733 εγκρίνεται. 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 219 Για τη 218 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 38-22. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 19 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 20 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ κατά αποχές Συγγνώμη, αλλά εγώ στο δικό μου τον κατάλογο ψηφοφορίας δεν έχει προβλεφθεί χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 262 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Διακόπτουμε την ψηφοφορία. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Χόουιτ. An oral amendment. sir. Με συγχωρείτε. Όχι χωριστή ψηφορία. Πρόκειται για σοσιαλιστική τροπολογία. Θέλουμε να βγει λέξη unlawful παρανόμως στα αγγλικά. Κατά τα άλλα, το κείμενο παραμένει ως έχει. Τροπολογία δηλαδή, αλλαγή πάνω στην δική μας τροπολογία. Να βγει η λέξη unlawful. Κατά τα άλλα, η τροπολογία παραμένει ως έχει. Λοιπόν, γιατί όχι, Χρειάζονται όμω δύο ψηφορίες τώρα. Μία με τη λέξη και μία χωρίς τη λέξη. Η πρώτη ψηφορία αφορά το κείμενο όσο έχει, το κείμενο της τροπολογίας, χωρίς την λέξη unlawful. Ψηφίζουμε λοιπόν επί του κειμένου χωρίς, επαναλαμβάνω, χωρίς τη λέξη unlawful. Πρώτη ψηφορία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το κείμενο. το κείμενο με τη λέξη unlawful. Ψηφίζουμε λοιπόν επί, ε, είναι το δεύτερο ρυθμό τη χωριστής ψηφοφορίας. Υπέρ. Κατά. Ωραία, απορρίπτεται. Συμβιβασμό 24. Υπέρ. Ο κύριο Λάσλορ. Μισό λεπτό πρέπει να επαναληφθεί το κείμενο. Καλή... Είναι η 24, μισό, λεπτό. Μας δόθηκε πριν από λίγα λεπτά, αλλά ήδη περιέχεται στον κατάλογο. Καλεί την κίνηση της Κούβας, όχι απλώ να ε, εξορίσει, λέει, τους πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά να τους δώσει την δυνατότητα να ταξιδεύουν στην Κούβα χωρίς να συλλαμβάνονται. Δεν βγαίνει νόημα από το κείμενο. Ε, προφανώς ε, οι αγγλόφωνοι εδώ θα μας διορθώσουν, αλλά το κείμενο προφανώς δεν βγάζει νόημα. Ελπιδοφόρο είναι αυτό. Λοιπόν, λίγα λεπτά, σας παρακαλώ. Επί του ιδίου και πολύ απλό. Καλή την κυβέρνηση της Κούβας να μην εξορίζει προφανώ. και να του δίνει ευκαιρία, την ελευθερία να ταξιδεύουν και να επιστρέφουν στην Κούβα χωρί να συλλαμβάνονται. Αυτό είναι η σωστή διατύπωση. Να μην εξορίζει. Καλείται να μην εξορίζει. Κάτι άλλο, αλλά για τα πρακτικά. Πρόκειται για νέο συμβασμό. Ψηφίζουμε ουσιαστικά επί του νέου συμβασμού, απλώς για τα πρακτικά να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι ψηφίζουμε επί διαφορετικού συμβασμού σε σχέση με αυτόν που συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Και ευχαριστώ ε, τους συνάδελφους που μας βοήθησαν να καταλήξουμε στην αυτή πρόταση. Ο κύριος Αλαφράγκα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να πούμε την αλήθεια, ο κύριος Λάμστορ έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά εμείς ψηφίσαμε το δεύτερο τμήμα της, τροπολογίας 262 και εδώ είχαμε και την, ε, την ε, συμβιβαστική τροπολογία της εισηγήτριας που ακύρωνε την τροπολογία του κυρίου Μπιόλς και πολύ καλοπροαίρετα ο κύριος Λάνσδορφ ε, όρμησε αυθορμήτως να μας αποδείξει την αντίφαση μεταξύ των δύο. Εγώ λέω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ε, να ψηφίσουμε την 24, τη συμβιβαστική δηλαδή και μετά να καταπέσει αυτή του κυρίου Ομπιόλ και τελείωσε. Εντάξει. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 24. Ο κύριος Χόουιτς θέλει το λόγο πάλι κύριος Σλαφράγκας με παρεξήγησε. Λέω ότι έχουμε διαφορετικό συμβασμό σε σχέση με τις κυρίες Αντεκίνη και αφορά τις δύο πρώτες γραμμές και μόνο και όχι ε, για το κείμενο το οποίο σχολήσε ο κ. Λάμπτροφ. Ε, πρόκειται για παρεξήγηση. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Η 2.36 καταπίπτει, γιατί η κυρία Αντρική είναι ευγενικά ενσωμάτωσε κάποιο από αυτό το κείμενο στη δική της τροπολογία και έτσι καταπιπτεί η άλλη. Μετά από μία ταπεινή ε, σκέψη να βγάλουμε δηλαδή το πείρμα Μέριλι από το κείμενο τελειώνει υπόθεση. το απλώς δηλαδή να βγάλουμε. Έχετε δίκιο, πρέπει να φύγει το Μιρλή, αλλά ο συνάδελφος έδωσε τη σωστή διατύπωση. Το δεύτερο μισό πρέπει να λέει και να τους δίνει την δυνατότητα να ταξιδεύουν και να επανέρχονται στην Κούβα χωρίς να συλλαμβάνονται. Για να βγάζει νόημα το κείμενο. Αυτή είναι η διατύπωση επί της οποίας πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, ωραία, άμα συμφωνούμε, έξω το Μέρλι, έξω το Απλός και τα βρήκαμε λοιπόν επιτέλους 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 278 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 279 υπέρ, κατά, αποχές, δεν το είδα. Η ηλεκτρονικά λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη 279. Πέρας της ψηφοφορίας. 27-23 εγκρίνεται. 280 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 281 αποσύρθηκε. 27 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 289 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 292 και 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 296 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 298 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 299 υπέρ. Κατά δεν το αυτό πάλι. Πάλι αφαιρεθήκαμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 299. Λέτε να προχωράω πολύ γρήγορα, λέει ο πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίες, η 29 29-25 απορρίπτεται 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 303 υπέρ Αχα, δεν πέρασε, είναι σωστά. Λοιπόν, 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 30 40 30, 30 διορθώνει το πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 307 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές αμφίβολο. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά και ελέγχω την 307. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 45-8. Όλοι ήταν υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία για την 308. Αρχίζει η ψηφοφορία. <coughs> Πέρας ψηφοφορίας 28-25 αρχίζει η ψηφοφορία για την 309 πάντα ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Το ίδιο έχουμε. 310 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 31 του εισηγητή. 316 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 317 και 18 μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 322 υπέρ κατά εγκρίνεται. 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα έλεγα λοιπόν τώρα για να τα απλουστεύσουμε τα πράγματα, να ψηφίσουμε unblock τις 324, 25, 26 και 27. Συμφωνείτε? Ναι? Α, ένας φτάνει, ωραία. Όχι. Ας δουλέψουμε τότε. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 327 υπέρ κατά εγκρίνεται 329 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 330 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 331 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 332 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 334 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 335 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 336 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα απορρίφθηκε να το ελέγξουμε όμως αρχίζει η ψηφοφορία για την 336. Ένα σωρό κόσμος δεν ψηφίζει. Για μία ψήφο απορρίπτεται. 25-24. 337 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 338 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 348 χωριστά λοιπόν πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 348, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Η 24 με 23 λοιπόν απορρίπτεται. 349 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 350 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 358 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 359 υπέρ κατά απορρίπτεται 360 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 361 υπέρ κατά εγκρίνεται 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 363 υπέρ κατά οι σοσιαλιστές ζητάνε να ψηφίσουμε ονομαστικά την 362. Η 362 λοιπόν ηλεκτρονικός Πέρες ψηφοφορίες. ψηφοφορίας. 18-32 εγκρίνεται. 363 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 364 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 367 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 371 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 372 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 374 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 375 υπέρ κατά εγκρίνεται 376 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 380 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 381 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 382 υπέρ κατά εγκρίνεται. 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 384 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 385 Ζητεί το λόγο η εισηγήτρια και της τον δίνουμε. Η κυρία Αντρική είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμβιβασμός 385. Ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα, διευκρινίσαμε κάποια πράγματα και το κείμενο άλλαξε ε, μάλλον το κείμενο λέει κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη στο Κογκρέσο το νομοσχέδιο ενώ το νομοσχέδιο και το ελέγξαμε με την πρεσβεία έχει ήδη υποβληθεί κατατηθεί στο Κογκρέσο και τώρα λέμε χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Μεξικού την καταπολέμηση του οργανωμένου ε, εγκλήματος και το νομοσχέδιο που έχει σαν στόχο να ε, ε, μεταρρυθμίσει κτλ. Ε, Συγγνώμη κύριε Αντρικίνη, μπορείτε να μας να επαναλάβετε αυτά που είπατε, τι θέλετε δηλαδή. Μάλλον διαβάστε το το καινούριο κείμενο. Ναι, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Μεξικού ναι, για τον αγώνα κατά της, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου ε, εγκλήματος και το νομοσχέδιο το οποίο έχει σαν στόχο τη μεταρρύθμιση της ε, στρατιωτικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει προσπευ... όλα αυτά να θεωρηθούν σαν ευκαιρίες για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει καλός, λέει ο πρόεδρος. Υπάρχει κανείς ε, που έχει ένσταση, αντίρρηση. Οκ. Okay. Λοιπόν, ψηφίζουμε 3.85 όπως το παρουσίασε η συγγήτρια. Παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.89. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 393 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 394 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 395 94 μάλλον έλεγχος ηλεκτρονική ψηφοφορία επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την 394 Chiusa la Πέρα τη ψηφοφορία. 25 κατά 23 υπέρ απορρίπτεται. 3,95 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβεβασμός 36. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3,96. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται 404 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 405 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 406 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 407 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 409 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 410 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 411 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 412 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 413 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 414 υπέρ κατά δεν είμαι σίγουρος. Ψηφίζουμε την 414 Ο κύριος Βέμπερ. Η κυρία Βέμπερ στην ε, λίστα λέει ότι μπορεί να αναδιατυπωθεί. Ρωτώ, έγινε αναδιατύπωση. Μεταξύ του Decides και Reconsider υπάρχει μεγάλη διαφορά κατά με. Ωραία, θα το ξεκαθαρίσουμε αμέσω. Να ελέγξει η γραμματεία το κείμενο. Mr. Chairman, it's your amendment. Πρόεδρε, δική σας ε, τροπολογία είναι αυτή. Ε, δεν τις θυμάμαι κιόλας απ' έξω, λέει ο πρόεδρος. E il testo della sulla lista di voto è quello Λοιπόν, ο Ρινάλντι δεν είναι εδώ. Αλλά εγώ είμαι υπέρ αυτής της διατύπωσης. Ωραία, ας ψηφίσουμε. 414, aperta la votazione. Λοιπόν, 414 αρχίζει η ψηφοφορία. Απέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 21 κατά. 415 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 416 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 417 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 418 υπέρ, κατά, αποχές, θα έλεγα ότι απορρίπτεται. 420 υπέρ. Α, δεν είναι ναι, δίκιο, έχετε. 419 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 420 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 421 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 422 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε λοιπόν το 15 ηλεκτρονικά. Chiusa la votazione elettronica sul 15. 39. Πέρας κατά 11 υπέρ. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 18 17 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 17. Chiusa la votazione. υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. 18 υπέρ. Ο κύριος Χάουιτ. Δεν είχα μετάφραση για ένα λεπτάκι. Ε, τέλος πάντων, ε, δεν ξέρω αν λειτουργεί τώρα η αγγλική μετάφραση. Εντάξει. Η 18 έλεγα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 27 a favore 23 contari approvato Εγκρίνεται 27-23. 23 λοιπόν τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 η ηλεκτρονικά την 26 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η 29 όχι, 19 ναι απορρίπτεται, η 27 υπέρ. Κατά αποχές. Εμένα μου φαίνεται ότι εγκρίθηκε, να ξεγκρίθηκε. Η 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ να ελέγξουμε την 28 Η 28 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται 25, ναι, 27 όχι, 31 ψηφίζουμε. 29, 29 λάθος, δεν πέρασε, σωστά, 29. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 31, 31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 32 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται,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 12 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και επιτέλους ηλεκτρονική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Imperitura gloria στην αυτοκράτηρα αντρική είναι πέρασε ομόφωνα η έκθεση. Λοιπόν, διακοπή μέχρι τον Επίτροπο. Όχι, όχι, όχι, ο Αυτοκράτορ Παντζέρη θα είναι τώρα. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio alla nostra seconda parte della sessione. Προχωράμε τώρα λοιπόν στην έκθεση του κυρίου Παντζέρη, Προέδρου της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Μαγκρέπ και της κυρίας Γκόμες που είναι η συγγήτρια για τις διαπραγματεύσεις σε μια συμφωνία πλαίσιο για τη Λιβύη μετά από την επίσκεψη στη Λιβύη στις 5 Νοεμβρίου. Όπως ξέρετε οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης είναι, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. Ο κύριος Παντζέρη ανέπτυξε πολλές επαφές ε, αυτού του τύπου με την αντιπροσωπεία του και μερικώς ε, πληροφορηθήκαμε για τις ε, διαπραγματεύσεις και την ολοκλήρωση της συμφωνίας πλαίσιο με τη Λιβύη. Να σας πω όμως τους εισηγητές πριν δώσω το λόγο ότι είχαμε επαφές με τον ε, ύπατο εκπρόσωπο στον οποίο ανέφερα ότι είχαμε δυσκολίες ε, για την πρόσβαση στα διαπραγματευτικά ε, έγγραφα. Είχα προφορικές απαντήσεις και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε για τη Λιβύη είχα την έκπληξη ότι ο πληροφορήθηκαν ότι το αίτημα αντί να το υποβάλουμε στην το πρόσωπο έπρεπε να την είχαμε στείλει στη Βελγική Κορεπέρ, δηλαδή στη Βελγική Προεδρία. Καλέσαμε λοιπόν έναν εκπρόσωπο της Βελγικής Προεδρίας για να μας πει τα σχετικά με την απόφαση η οποία ελήφθη. Αυτά εισαγωγικά. Και χωρίς άλλες καθυστερήσεις δίνω το λόγο στον κύριο Παντζέρη για να μας πει τα σχετικά. Πέντε χρόνια δεν έλειπε από τη Λιβύη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπροσωπεία μας είχε δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, να ενισχύσει τις σχέσεις με αυτή τη χώρα που θεωρούμε στρατηγικό συνομιλητή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση, την ενέργεια και επίσης ως παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας στην Αφρική. Ο ρόλος τώρα του Κοινοβουλίου αναβαθμίζεται λόγω της ε, Λισαβόνας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέσαμε και στους συνομιλητές μας ε, διάφορες ερωτήσεις που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Η φάση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης, διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, προγράμματα στον τομέα της υγείας, η υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετοχή της Λιβύης ε, στα προγράμματα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ε, και τη διαχείριση των υδάτων και την ε, καθαρή ενέργεια. Επίσης για τη σύμβαση της Γενέβης του 1951 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μορατόριο στη Λιβύη για την θανατική ποινή. Βέβαια είχαμε μερικά οργανωτικά προβλήματα τα οποία μας δημιούργησαν οι οι αρχές της Λιβύης και μας άλλαξε τα προγράμματα από την πρώτη ημέρα, μας ενόχλησε αυτό και είχαμε και πολλές πολεμικές, ίσως και πρόορες, γιατί μετά η κατάσταση διορθώθηκε <coughs> και διαπιστώσαμε ποια είναι η κατάσταση στη χώρα αυτή. Και λόγω της επίσκεψης που κάναμε σε ορισμένες σημαντικές υποδομές στη Βενγάζη και οι πολιτικές μας συναντήσεις στην Τρίπολη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μία πολιτική εκτίμηση. Υπάρχει μία διαλεκτική μεταξύ συντηρητικών ε, και νεοτεριστών και στις καθημερινές σχέσεις το βλέπουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι λοιπόν στατικά τα πράγματα στη Λιβύη. Πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση από κοντά γιατί αυτό θα έχει επιπτώσεις και εσωτερικά και διεθνώς και επίσης και σε αλλαγές στην λιβική νομενκλατούρα που μπορεί να αλλάξει. Τώρα υπάρχει, το να πούμε ότι υπάρχει μια ευθυγράμμιση σε αυτή τη συζήτηση δεν είναι, θα, θα ήταν άτοπο. Αλλά η διαδικασία είναι ενδιαφέρουσα και θα έπρεπε να την παρακολουθήσουμε. Αυτή την αίσθηση την είχαμε στις επαφές μας στην Τρυπολίτιδα και στην ε, Βενγάζη και σας τα μοιράσαμε και γραπτά αυτά στο έγγραφό μας όπου ο, ο γραμματέας γενικών υποθέσεων της Επιτροπής ε, της Εθνοσυνέλευσης του Λαού δεσμεύτηκε να μας δώσει ένα συγκεκριμένο έγγραφο που να κάνει αναφορά της κατάστασης στη Λιβύη και θα είναι ίσως η μόνη χώρα του, του μετά το Μαρόκο που μας δίνει μια τέτοια έκθεση. Υπάρχουν φυσικά προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμείς μπορούμε να θεωρήσουμε ως άνοιγμα ε, τις δηλώσεις που μας έγιναν να συμμετέχει η Λιβύη στη Συμφωνία του της Γενέβης του 51 για τους πρόσφυγες. Όπως επίσης ε, ε, και το άνοιγμα γραφείου και με το άνοιγμα γραφείων της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες ε, φαίνεται να μας δείχνουν μια καλή θέληση. Θεωρούμε λοιπόν ότι είμαστε ικανοποιημένοι γιατί μπορεί να ξεκινήσει μια νέα φάση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Λιβύης και επιβάλλει την παρουσία του δυναμικά το Κοινοβούλιο την παρουσία του στη Λιβύη. Επίσης θα χρειαστεί κάποια στιγμή να ανοίξουμε και μία αντιπροσωπεία στη Λιβύη για να συνοδεύσουμε όλες τις διαπραγματεύσεις που ε, τρέχουν σήμερα. Εμείς ε, πιστεύουμε στο διάλογο με τη Λιβύη και η υπογραφή του συμφώνου πλαισί, της συμφωνίας πλαίσιο πρέπει να λάβουν υπόψη αυτό το πλαίσιο και αυτούς τους όρους. Θεωρούμε λοιπόν ότι μετά από αυτή την επίσκεψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει μια πρώτη σύσταση στο Συμβούλιο ε, χρήσιμη για να ενσωματώσει τις κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, για τη συμφωνία πλαίσιο. Τώρα, σύντομα συμπερασματικά σχόλια. Ευχαριστούμε τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λείπει πάντως μια συνεργεία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να θεωρεί ως βοήθεια τη δουλειά του Κοινοβουλίου και όχι ως εμπόδιο ή ενόχληση. Δεύτερον, πρέπει να εξηγήσουμε σωστά και ένα περισσότερο το νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη συνθήκη. Αυτό ισχύει και για τη Λιβύη, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους. Είναι ένας όρος συνεκονών. Ε, γιατί είμαστε πλέον θεμελιώδεις συνομιλητές. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν τη γραμματεία της Επιτροπής για την εξαιρετική της δουλειά και στην προετοιμασία αλλά και στην παρουσία στην ε, Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχαριστίες ε, για, εξωτερική, για όλη την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που ξεχάστηκαν βέβαια αλλά τις, ε, τους δεχόμαστε. Η κυρία Γκόμες. Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι η Λιβύη πραγματικά έχει μεγάλη στρατηγική σημασία για την Ευρώπη. Κάποια από τα, αρκετά από τα κράτη-μέλη μας έχουν ε, πολύ στενές και διε, με τη Λιβύη που επεκτείνονται κιόλα. βεβαίω είναι δικτατορία η Λιβύη, από πολιτικής απόψεως αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα, αλλά από οικονομική και κοινωνική άποψη ε, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, κακά γιατί υπάρχει σχετικά δίκαιη κατανομή των, των εσόδων από το πετρέλαιο. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον για μένα το γεγονός ότι στην επίσκεψη μας ε, μπορέσαμε να θέσουμε όλα τα θέματα που σχετιζόταν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κανείς δεν μας αρνήθηκε μια απάντηση και όπως είπε και ο κύριος Παντσέρη ήταν πάρα πολύ καλή η συνάντηση και είχαμε υψηλό επίπεδο συνομιλητές ε, αντίστοιχους ας πούμε με τον πρόεδρο της Βουλής στις δικές μας χώρες. Δε, όπως είπε και ο Αντώνιο Παντσέρη δέχθηκε και η Λιβύη το, ότι υπάρχει πιθανότητα να συμπογράψει, συμμετάσχει στην συνθήκη για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρουμε από εκεί και πέρα ότι και ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι στη Γενέβη λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις και συνομιλίες μεταξύ Λιβύης και είπα της αρμοστίας για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί και έχει μεγάλη σημασία από εκεί και πέρα η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει τη Λιβύη, δεν μπορεί να είναι αδιάφορη στην οποιαδήποτε ανάπτυξη και εξέλιξη της Λιβύης. Βεβαίως μπορεί να κάνει λάθη η Λιβύη, αλλά το θέμα δεν είναι... Η, την σήμερα ημέρα πρέπει να συνάπτουμε σχέσεις, όχι να απομακρύνουμε και να απομονώνουμε άλλους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη και εντονότερη παρουσία στη Λιβύη. Να θα μπορούσε να ανοίξει ο πολιτικός χώρος για επαφές με τη Λιβύη όπως γίνεται με το σχέδιο δράσης Μπενγκάζη για να δημιουργηθεί κέντρο αριστείας κατά του AIDS στην ε, Μπενγκάζη παρεπιπτόντως φαίνεται ότι αυτό το κέντρο έχει τεράστιες, ε, τεράστια, πολύ καλά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι θέλουν να επεκτείνουν τώρα το κέντρο ε, και σε άλλες μολυσματικές ασθένειες, λοιμώξεις κτλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, υπάρχει βέβαια η συμφωνία πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να αναθεωρηθεί η συμφωνία αυτή Αμέσω θα πρέπει κατά την άποψή μου να στείλουμε μήνυμα στο Συμβούλιο ζητώντα να αναθεωρηθούν οι όροι διαπραγμάτευσης. Εκείνο το οποίο είναι απολύτως απαράδεκτο είναι ότι το Συμβούλιο προσπαθεί μέσω της Κομισιόν να φτάσει σε μια συμφωνία επανεισδοχής. Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο. Μιλάμε για μια δικτατορία, μιλάμε για μια χώρα που μπορεί τώρα να είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών για, όσον αφορά τα ανθρώπινα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Ε, συμφωνία επανεισδοχής με τη Λιβύη, απαράδεκτο. Και ούτω ή άλλω και η Λιβύη η Λίβοι δεν θα το δοχόντουσαν ποτέ. Το Συμβούλιο, κυρία Άστον, δεν μας αποκάλυψε ακόμη τους όρους της ε, διαπραγμάτευσης αλλά οι Λίβοι μας είπαν ήδη ότι ζητείτε κάτι τέτοιο, συμφωνία επανεισδοχής από τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, εδώ πρέπει να προσέξουμε. Επίσης θα πρέπει να επιμείνουμε να ε, συμμετάσχει η Λιβύη ε, στις ε, συμβάσεις και συνθήκες για τους πρόσφυγες. Ε, αυτό θα ήταν πολύ καλό για όλους μας και εκείνο που προσπαθούμε όλοι μας να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τους μετανάστες και τους ετούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Γιατί λοιπόν ε, να μην βοηθήσει και Λιβύη. Θα ήταν πολύ καλό επίσης το Συμβούλιο να προσφέρει ένα κάποιο πρόγραμμα επανακατάστασης για τους ετούντες άσυλο και για τους πρόσφυγες. Επίσης θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόγραμμα παροχή συμβουλών και τα λοιπά και θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε και εμείς να ομισθούμε ένα μέρος του βάρους. Αν άλλη μεριά υπάρχει και βεβαίως και νόμιμη μετανάστευση. Πρέπει να αντιλάβουμε υπόψη διότι οι μεταναστευτικές ροές που περνούν αυτή τη στιγμή από τη Λιβύη ε, ε, ε, σχετίζονται όπως και σε άλλα μέρη ε, με, την, με το λαθρεμπόριο ανθρωπίνων όντων. Λοιπόν, θα πρέπει να επιμείνουμε. Θα πρέπει να μας δοθούν στοιχεία, πληροφορίες για αυτό το θέμα, για αυτούς που πρόσφατα εξετελέστησαν ε, θανατική ποινή και τα λοιπά. Ε, και είναι, θα ήταν πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και την κοινωνία των πολιτών. Φαίνεται βέβαια να γίνονται κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, να υπάρχουν κάποιες κινήσεις για να βγουν από την απομόνωση οι Λίβοι. Οπότε θα πρέπει να τα ενισχύσουμε αυτά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε επίσης προγράμματα για τα δικαιώματα των γυναικών, τέτοιου είδους προγράμματα. Και θα πρέπει να πιέσουμε η Λιβύη να συμμετάσχει σε μια περιφερειακή ένωση αν θέλετε αναπτυξιακή αυτό νομίζω ότι το θέλουν και οι Λίβοι Α, για το περιβάλλον επίσης, προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές αλλαγές. Η Λιβύη αυτή τη στιγμή είναι κύρια αιτία για κάποια περιβαλλοντικό προγράμματα της περιοχής αυτής για την α, απερίμωση και την έλλειψη ύδατος σπάνι ύδατος παραδείγματος χάρη οπότε καλό θα ήταν να τους πιέσουμε τους Λίβιους να συμμετάσχουν σε κάποια τοπική ε, περιφερειακή ένωση που θα δουλεύει για αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε και το σύστημα των θεωρήσεων βεβαίω της βίζας. Ε, είναι σημαντικό το θέμα και για τους Λίβιους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία είναι επιφυλακτικά. Δεν ξεχνάμε το Λόκερμπι, δεν ξεχνάμε τη δίσκο στο Βερολίνο το σύστημα βίζας Schengen θα μπορούσε όμως να εφαρμοστεί και μάλιστα γρήγορα. Αυτό κατ' εμέ είναι εφικτό. Και αν γινόταν κάτι τέτοιο θα καθησύχαζε κάποιους, θα διασκέδαζε κάποιους φόβους και κάποιες ανησυχίες. στεναχωρήθηκα που η συνάδελφος Αλφάνελ βγήκε από τη Λιβύη και έκανε τις δηλώσεις που έκανε χωρίς να έχει παρακολουθήσει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αυτά που είπε στις δηλώσεις τις αντιστοιχούν με αυτά που είδαμε εμείς στη δική μας την επίσκεψη. Και θα της το πω, δεν ξέρω που είναι αν είναι παρούσα εδώ, αλλά όταν τη δω θα της πω ότι διαφωνώ με αυτά που είπε. Κακώς έδρασε με αυτόν τον τρόπο κατά την άποψή μου. Το είπα και το επαναλαμβάνω αυτό. Επίσης, καλό θα ήταν να κινηθούμε γρήγορα, να περάσουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Άστον, διότι τα φτάνουν στην τελική τους φάση οι διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι ως το δυνατόν πιο γρήγορα θα πρέπει να κινηθούμε για να εγκρίνουμε και ένα ψήφισμα με συγκεκριμένε συστάσει. Και βέβαια θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα πράγματα. Engagement, συμμετοχή και στενή σχέση είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, όχι απομόνωση. Ο κύριος Γιακολίνο, μέλος της Επιτροπής. Συμμετείχα λοιπόν κι εγώ σε αυτήν την αντιπροσωπεία. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε ιδιαίτερα χρήσιμες συναντήσεις, κυρίως την τελευταία μέρα που εγώ δεν μπορούσα να συμμετέχω, αλλά και τις προηγούμενες είχαμε πολύ καλές συναντήσεις. Επρόκειτο περί γενικού και προσωπικού εμπλωτισμού γνώσεων είχαμε κίνητρα, μας δόθηκαν κίνητρα θετικά και για την ερίσματα πολύ θετικά για να προχωρήσουμε Βέβαια απέχει παρασάγκαση Λιβύη από τη δυτική πραγματικότητα. Αλλά είδαμε ότι υπάρχει ένα πυρήνα υποδομών και σχεδίων που ε, εξελίσσονται και πρέπει να ολοκληρωθούν, πρέπει να λάβει υπόψη η Κομισιόν βέβαια στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων ορισμένα στοιχεία Εμείς θα τα υποστηρίξουμε, θα, θα υποστηρίξουμε βέβαια, αλλά μην αγνοήσουμε το προφίλ που αφορά στην Μεσόγειο. Εκείνο το, το, το στοιχείο εκείνο το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε όταν μιλάμε για Μεσόγειο. Η αλληλεία. Ας πούμε στον κόλπο της Ήρτης υπάρχει πρόβλημα ε, ε, ξέρουν πάρα πολύ καλά οι λιβικές αρχές. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η πρόσφατη συμφωνία με την Ιταλία που είναι παραδειγματική και για τη διακίνηση των, ε, και για τον έλεγχο των μεταναστών κτλ. Πρέπει να βγάλουμε τη Λιβύη από το περιθώριό της Πρέπει λοιπόν σίγουρα να τις ανοίξουμε τις πόρτες στη Λιβύη, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και τη σωματεμπορία και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την τρομοκρατία. Συμφωνώ με τον Παντζέρη που λέει ότι πρέπει να εκφράσουμε εμείς προς το Συμβούλιο τη βούλησή μας να υπάρξει συμφωνία πλαίσιο και σύντομα μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο, κύριο Σαρλάκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Παντζέρη και την αντιπροσωπεία μας στη Λιβύη. Καταρχήν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, διότι έδειξαν τι μπορεί να κάνει αυτό το Κοινοβούλιο. Να καλύψετε δηλαδή ένα κενό στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Αναλάβαμε πρωτοβουλία. Είμαστε σε διάλογο με μια χώρα σημαντική για την Ευρώπη αλλά και για πολλά κρατημέλη. Και δείξαμε ότι αυτή η μέθοδος αποδίδει. Ο διάλογος δηλαδή και η συνεργασία. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύστημα, όταν δηλαδή δρά, όταν ενεργεί σύμφωνα με τον βαθύτερο σκοπό της. Και διαφοροποιούμενη έτσι με την αμερικανική πρακτική έναντι χώρων όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε, κατάρρεσαν την Λιβύη μεταξύ των χωρών παρίες του άξονα του κακού Όπω λέγαμε πριν λίγα χρόνια. Εμείς δεν ε, στενιστήκαμε αυτήν την ε, προσέγγιση, η οποία είχε αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση της Λιβύης, η οποία από απελπισία, μην έχοντα τίποτα άλλο να κάνει, υποστήριξε την δημοκρατία και προσπάθησε να εξασφαλίσει και όπλα μαζικής καταστροφής. Το γεγονό ότι η Λιβύη σε κάποιο βαθμό υιοθέτησε την ευρωπαϊκή προσέγγιση είχε ακριβώς το αποτέλεσμα να αφοπλιστεί και να εγκαταλείψει και τις ε, προνομιούχες σχέσεις με την ε, τρομοκρατία και την διεθνή βία. Και αυτό ακριβώ αποτελεί τεράστια επιτυχία της διεθνούς κοινότητας και για την ευρωπαϊκή μέθοδο, αν θέλετε, του εξωτερική πολιτική. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ε, το Ιράν για παράδειγμα. Πιστεύω ότι η ειρηνική προσέγγιση θα έχει τελικό το πάνω χέρι. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο εν τέλει πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε σε αυτή την κατεύθυνση, θέλοντας δεδομένο ότι δυστυχώ η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν ηγούνται δυστυχώ αυτή τη ε, προσπάθεια. Όμω το σύστημα αυτό, το Κοινοβουλίο αναλαμβάνει τι ευθύνε του και ανοίγει νέους δρόμους στην εξωτερική πολιτική. Η σχέση βεβαίως με την Λιβύη ξεκίνησε χάρη στις προσπάθειες του κ. Πρόντι που άλλαξε ριζικά την προηγούμενη προσέγγιση. Η ιταλική εμπειρία των σχέσεων με τη Λιβύη είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ευθυγραμμίζεται θα έλεγα συνάδει με την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια στην Ιταλία, στην πολιτική εναντί τη Λιβύη, μεταξύ των ε, αριστερών και των δεξιών κυβερνήσεων, των κεντροδεξιών κυβερνήσεων. Κάτι το οποίο είχε και πάλι τα αποτελέσματα στον τομέα τη ε, μετανάστευση, τη ενεργειακή συνεργασία. και αυτό με τη σειρά του είναι και πάλι πολύ σημαντικό για την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Λιβύα. Στη Λιβύη, με συγχωρείτε. Οι κυρώσει και οι μεγαλιστομίε δεν αποδίδουν. Η δική μα μέθοδο είναι η κατάλληλη μέθοδο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Το να κατηγορούμε ασύστολα την Λιβύη δεν μα κάνει καλύτερου, ούτε βελτιώνει την κατάσταση για μα. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λιβύη, να βελτιώσουμε τα τη κοινωνία των πολιτών, πρέπει να συνεχίσουμε στον δρόμο που έχουμε ακολουθήσει ω σήμερα, μακριά από κυρώσει και ακραίε αντιμετωπίσει. Η δική μα μέθοδο, η δική μα προσέγγιση θα λύσει τα προβλήματα, μακριά από εντάσει. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα στην ίδια κατεύθυνση και να δείξουμε στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό σύστημα το δρόμο. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο έχει και άλλα μέσα στα χέρια του, πέρα από την Συμφωνία Πλαίσιο και άλλες ε, συμφωνίες και θα συνεχίσει, πιστεύω, να δίνει το παράδειγμα στον τομέα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάκη. Ο κύριος Λάνστορφ. Πρόεδρε. διερωτήσεις. Ε, εκπλήττουμε θετικά, γιατί προς το παρόν είχα δει μόνο το email Ερφάνο ε, και είχα αρχίσει να λαμβάνω αντιφατικά μηνύματα. Αν και συμφωνώ ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τη Λιβύη. Έχω πάντω κάποιε ερωτήσει και κάποια σχόλια που θέλω να διατυπώσω. Πρώτον, ποιο είναι το περιεχόμενο τη συμφωνία πλαίσιο, τι πρέπει να λέει αυτή η συμφωνία, να το συμφωνήσουμε αυτό εδώ. Δεύτερον, α μην έχουμε ψευδεστήσει, η Ανά Γκόμε ήταν, είπε τα σιγά σιγά και της Καρσκάφη όταν μα είπε ότι η Λιβύη είναι δικτατορία και περί αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Συνεπώ. Ας μην, έχουμε, ας μην διατηρούμε φρούδες ελπίδε. Α θυμηθούμε πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Ελβετία και Λιβύη για κάποιο χρονικό διάστημα εξαιτία ενό ε, επεισοδίου το οποίο υποτίθεται ότι αποτελούσε ε, μορφή κατά της ε, οικογένειας του δικτάτορα. Είχαμε συλλήψεις ο Μύρον, πράγματα απαράδεκτα για μια χώρα που είναι υποτίθεται στρατηγική σημασία για την ε, Ευρώπη. Βεβαίω ε, είναι, συνεχίζει να είναι σημαντική. Τρίτον, η επανεισδοχή. Δεν νομίζω ότι η συμφωνία επανεισδοχή πρέπει να είναι τμήμα μια γενικότερη συμφωνία, γιατί δεν εξάγει μόνο μετανάστε η Λιβύη, αλλά είναι και σημείο διέλευση το να ζητήσουμε λοιπόν κάτι τέτοιο, μια συμφωνία επανεισδοχής, δεν μου φαίνεται τόσο ακραίο και εξαιρετικά φιλόδοξο. από την άλλη μεριά αισθάνομαι σε ταινία του Μπουνιουέλ. Διότι συζητούμε τη συνεργασία με τον Καντάφη στο πλαίσιο μια ε, συμφωνία πλαίσιο, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό βεβαίω, αλλά όταν ε, έρχεται η στιγμή να συζητήσουμε κάποια μικρή αναβαθμίση των σχέσεων μα με το Ισραήλ, ε, κολλάμε σε λεπτομέρειες όπως ε, η αμοιβαία αναγνώριση φαρμακευτικών προτύπων κλπ. Ναι λοιπόν στη συνεργασία, αυτή είναι η ευρωπαϊκή μέθοδος, η ευρωπαϊκή προσέγγιση, συμφωνώ με αυτό, αλλά αν είμαστε σε θέση να το καταφέρουμε αυτό με χώρες δύσκολε, χώρες δικτατορίε αν θέλετε, τότε θα έπρεπε πολλό μάλλον να πράξουμε το ίδιο με χώρε που είναι δημοκρατίες και που έχουν αποδείξει την διάθεσή τους να συνεργαστούν. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Λάστορφ. Βαρτζέτ. Oui, Monsieur le Président. Euh, je vais être assez rapide. Je voudrais... Πρόεδρε, θέλω να καταγγείλω το κλίμα σε αυτήν την Επιτροπή. Διότι δεν μου αρέσουν αυτά τα οποία άκουσα από συναδέλφους κυρίως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη συμφωνία πλαίσια με τη Λιβύη, και δεν συμβαίνει τίποτα. Τη στιγμή που ξέρουμε τι είναι αυτή η χώρα, η Αναγκόμες το είπε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι διακυβεύεται στις συνομιλίες για την Ιταλία. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις απειλές και τους κινδύνους που απειλούν μετανάστες ε, και κυρίως ετούντες ε, άσυλο. πιστεύω ότι πάμε να κάνουμε αυτό, ε, ακριβώς το αντίθετο αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε την Ευρώπη φρουρή και από την άλλη τους πολιτικούς στόχους, τους οικονομικού στόχους. Εγώ δεν μπορώ να σιωπήσω και να αγνοήσω την πραγματικότητα. Διαφωνώ με τα όσα ακούστηκαν. Για μένα δεν είναι δυνατόν να υπογράφουμε συμφωνίες τη στιγμή που πολύ βασικέ αρχέ των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν τηρούνται. Και δεν πιστεύω τι υποσχέσει των Λιβύων προκειμένου. Όπω είπε και ο συνάδελφο Λάνστορφ, ξέρουμε πολύ καλά που πηγαίνουν οι υποσχέσει τη Λιβύη και μάρτυρέ μα και οι Ελβετοί, οι οποίοι έχουν ήδη πήραν του θέματο. Ο εκπρόσωπος τη Κομισιόν, Δόκτωρ Μπρουνέη αν θέλει βεβαίω να σχολιάσει, εάν το επιθυμεί και μόνον. Καλησπέρα. Το μόνο το οποίο θα μπορούσα να παραλάβω ενώπιον σα σήμερα, μια που μου δίνετε τον λόγο, είναι πρώτον να σα ευχαριστήσω. Δεύτερον, η Κομισιόν είναι διερθυμένη να συνεχίσει την πολιτική καταρχήν που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να συνεχίσει δηλαδή την πολιτική προσέγγιση με την Λιβύη εδώ και αρκετό καιρό. Είμαστε υπέρ της, συνεργασίας, διότι υπάρχουν συμφέροντα μεταξύ Λιβύης και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διότι η σύμπραξη, η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε την κατάσταση, την πολιτική, την κοινωνική στη χώρα αυτή. Μια πολιτική η οποία βεβαίως πρέπει να συνάδει με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να προσθέσω επίση ότι η Κομισιόν σε ορισμένε χρονικές στιγμές διακινδύνευσε ε, για να προχωρήσουν οι σχέσεις αλλά και να αντιμετωπιστούν ε, καταστάσεις ε, ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος ε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο κοινωνικό ανακοινωθέν για την μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή απέδειξε ότι έχει τη διάθεση να συνεργαστεί επικοδομητικά με έναν εταίρο ο οποίος παραμένει κατά κοινή ομολογία δύσκολος. Όσον αφορά τώρα τι διαπραγματεύσει για την συμφωνία πλαίσιο, αυτό το οποίο σήμερα θα μπορούσα να σα πω είναι ότι ο επόμενο γύρο θα λάβει χώρα μεθαύριο στην Τρίπολη. Είναι μάλλον πρόωρο, θα είναι υπερβολικά πρόωρο, να προβλέψω την κατάληξη αυτών των διαπραγματεύσεων, οι οποίε, όπω πολλοί παρατήρησαν, παραμένουν δύσκολε τόσο για τα εμπορικά θέματα όσο όσον αφορά και την μετανάστευση και την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών των προσφύγων. Εμείς θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης από το, τα τέλη της εβδομάδας δηλαδή, ε, όπως άλλωστε το πράξαμε σε κάθε παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στους δύο εισηγητές, την κυρία Γκόμες και τον κύριο Παντζέρη για τα τελικά σχόλια. Πρόεδρε, συμφωνώ με τους συναδέλφους. Ναι, έχουμε να κάνουμε μία δικτατορία, όμως είναι μία δικτατορία στη γειτονιά μας και πρέπει να συνεργαστούμε για να μειώσουμε ακριβώς τις επιπτώσεις των πολιτικών ορισμένων κρατών μελών, κυρίως όσον αφορά την μετανάστευση. Αν αυτό δεν μπορέσουμε να το κάνουμε στο πλαίσιο μιας υποδιαπραγμάτευση συμφωνία, παρουσία και της υπατισαρμοστίας του ΟΗΕ για του πρόσφυγες, τότε θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο μας, να προστατεύσουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν πολύ δύσκολα στην Λιβύη. Πέρα από τους πρόσφυγες και τους ε, παρανομού μετανάστες, έχουμε και τις συνθήκε διαβίωσή του. Η Λιβύη δεν θεωρεί ότι έχει παρανομού μετανάστες, ε, θεωρεί ότι έχει προσκεκλημένους εργάτες. Και εκεί συμβαίνουν φοβερές διακρίσεις. Εμείς πρέπει να έχουμε παρουσία στην περιοχή. Πρέπει να διαδραματίσουμε ρόλο, να συλλέξουμε πληροφορίες και να προλάβουμε τα χειρότερα. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Κάποια κράτη-μέλη είναι ήδη εκεί και μάλιστα όχι όπως θα έπρεπε. Υπό τις λάθος προϋποθέσεις. Ας κάνουμε κάτι να βελτιώσουμε την κατάσταση. Από όσα είδα, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια σημάδια ανοίγματο. Κάτι κινείται. Η κοινωνία των πολιτών ακολουθεί τα βήματά μας. Ας τη βοηθήσουμε. Υπάρχουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δύναμη, επεκτείνονται και αυτές πρέπει να τις βοηθήσουμε. Και στο κάτω-κάτω Κανείς δεν είναι τέλειος. Δεν μπορούμε να υπογράφουμε συμφωνίες μόνο με μη δικτατορίες. Και δεν το έχουμε πράξει ποτέ αυτό ούτως ή άλλως. Έχουμε συμφωνίες και με άλλες δικτατορίες. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Οπότε σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση εγώ τουλάχιστον είμαι απολύτως πεπισμένη ότι κάνουμε το σωστό. Η συμφωνία πλαίσιο θα έχει καλά αποτελέσματα και εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε αρμοδιότητα προκειμένου. Εμείς τους είπαμε, είπαμε του Λίβιου, όπω το είπε ο κ. Παντσέρη, ότι χωρίς εμάς συμφωνία δεν γίνεται. Λοιπόν, α εργαστούμε για μια καλύτερη εξέλιξη, για καλύτερε εξελίξει στην Λιβύη. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πεπισμένη. Ο κ. Παντζέρη. Non c'è da parte nostra... Θέλω να διασφαλίσω ορισμένου ε, συνεδελφούς ότι δεν είμαστε καθόλου αφελείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ε, τι αντιμετωπίζουμε όταν συζητάμε με τις ε, λιβικές ε, αρχές. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ούτε μία συνέχεια ούτε και προβλεψιμότητα στη στάση των λιβικών αρχών. Εγώ λέω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο και τις σχέσεις μας και να θέτουμε τους δικούς μας όρους που είναι σαφείς και τους ανέφερε και η Άννα Δεν μπορούμε στρουθοκαμιλίζοντας να λύσουμε το πρόβλημα των προσφύγων και των μεταναστών. Σίγουρα καθησυχάζουμε τη συνείδησή μας αλλά δεν ε, παίζουμε το ρόλο μας ως βουλευτές ε, και δεν παίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ρόλο του. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερο κουράγιο, περισσότερος ενθουσιασμός και στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράγμα το οποίο πολλές φορές διαφεύγει και πρέπει να το τονίζουμε. Είναι σαφέστατα τα συμπεράσματα. Εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να διατυπώσουμε συστάσεις ε, στο Συμβούλιο ούτω ώστε η συμφωνία πλαίσιο να συμπεριλαμβάνει και τις δικές μας εκτιμήσεις. Σύμφωνοι λοιπόν για μια συμφωνία πλαίσιο αλλά και με τις δικές μας παρατηρήσεις. Σε ευχαριστώ λοιπόν όλους. Ε, θεωρούμε ολοκληρωμένη την συζήτηση με αυτό το τόσο με όλα αυτά τα αιτήματα που ε, διατύπωσαν οι συνάδελφοι, δηλαδή να υποβάλουμε εμεί μία σύσταση που να λέει ότι η συμφωνία με την Λιβύη πρέπει να εγγραφεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και να εκφράζονται σε αυτήν τη σύσταση όλα όσα μας αναφέρατε. Σας ευχαριστώ, διακόπτουμε για να ξαναρχίσουμε στις 6 με την ακρόαση του κυρίου Φούλε.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 Και εμείς αυτό αναρωτιόμαστε. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι τι. Αν πρόκειται, αν στη συνέντευξη τύπου λέει αυτά που θα έρθει να μας πει εμάς, τότε να πάμε σπίτι μας από τώρα. Ε. Δεν το δέχομαι αυτό να πει πρώτα στον τύπο τι είναι να πει. Μα αφού το επαληθεύσουμε βεβαίως, αυτό θα κάνουμε. Uh, Συμφωνώ ότι πράγματι αν τα ίδια πράγματα ανακοινωθούν δημοσία στο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, τότε δεν χρειάζεται να τα ξαναπεί εδώ και ο Επίτροπος. Η συνάντησή μας είναι για τις 6. Πιο μπροστά υπάρχει συνέντευξη τύπου. Όταν έρθει ο Επίτροπος να ρωτήσουμε αν έγινε συνέντευξη τύπου και με τι αντικείμενο. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιμείνουμε και να δημιουργήσουμε μεγάλο πρόβλημα λόγω αυτή, αυτού. Ναι, μου το επιβεβαίωσαν ότι ο κύριος Φίλε μετά από την ε, συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων έδωσε μία συνέντευξη τύπου «Ε, όταν θα έρθει εδώ θα του πούμε να μας αναφέρει τι είπε προηγουμένως στον τύπο αντί να μας τα πει σε εμάς που είμαστε και το αρμόδιο θεσμικό όργανο Bene colleghi, possiamo iniziare la nostra riunione. Il commissario Füle ci ha raggiunto. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ήρθε και ο Επίτροπος με τέσσερα λεπτά καθυστέρηση, ε, σπάνιο για την περίπτωσή του, γιατί πρόκειται για κάποιον που είναι πάρα πολύ ακριβής. Αλλά όπως συνέβη και στον Όμηρο λέει ο πρόεδρος εννοώντας τον Οδυσσέα, τον πήρε ο ύπνος. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω εδώ, ήρθε μάλλον να μας αναφέρει ο Επίτροπος, για τις ε, χώρες που πρόκειται να γίνουν μέλη, είναι ενδυνάμει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν προοπτικές ε, για τις διαπραγματεύσεις με την Κροατία, ε, με την ε, πρώην ε, δημοκρατία της, ε, Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, υπάρχουν οι ημερομηνίε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, τέλος πάντων υπάρχουν ένα σωρό πολύπλοκα σενάρια τα οποία θα μας αναφέρει εδώ ο Επίτροπος. Τώρα κύριε Επίτροπε βέβαια να σας πω, εσείς πάντα έχετε αυτή την ευαισθησία να άρχεστε εδώ να μας διηγήσετε όλα τα σενάρια. Αλλά σε αυτά τα λίγα λεπτά τα οποία μεσολάβησαν από το συμπέρασμα ε, ε, από την ολοκλήρωση μάλλον της ε, συνεδρίασής σας και της δικής μας συνάντησης, ορισμένοι συνάδελφοι διαπίστωσαν ότι αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων προχωρήσατε σε μια συνέντευξη τύπου. Πριν τα συζητήσετε τα πράγματα με εμά που είμαστε και το θεσμικό όργανο που έπρεπε να συζητηθούν όλα αυτά. Εγώ δεν είμαι κατά του γεγονότος ότι εσείς θα πρέπει να ανακοινώνετε αυτά τα οποία <coughs> αποφασίζονται στα δικά σας όργανα και στα πλαίσια του ρόλου σας και των ευθυνών σας. Αλλά ορισμένοι συνάδελφοι έθεσαν αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθα μας ε, εξηγήσετε, θα μας δώσετε μια απάντηση σε αυτό το λεπτό και κριτικό θέμα. Σας δίνω το λόγο λοιπόν αγαπητέ Επίτροπε. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ πρόκειται για το πρώτο πακέτο διεύρυνσης το δικό μου και γιατί το λέω έτσι, γιατί όταν θα παρουσιάσω το δεύτερο πακέτο διεύρυνσης ε, μπορεί να έρθω τρία λεπτά πιο πριν και γιατί μπορεί να μην ισχύουν οι ίδιες μοναδικές συνθήκες που ισχύουν σήμερα Δηλαδή, τι έγινε σήμερα η συνάντηση των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έγινε το πρωί όπως ήθιστε να γίνεται, αλλά άρχισε το, το μεσημέρι. Και με, άμα γινόταν το πρωί, αν είχε γίνει μάλλον το πρωί η συνάντηση, όπου μετά τις πρωινές συναντήσεις των Επιτρόπων έρχομαι κατευθείαν στο Κοινοβούλιο και μετά πάω στους δημοσιογράφους. Αλλά σήμερα τα πράγματα ήταν μοναδικά, ήταν διαφορετικά. Παρά όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ήταν μοναδικές, προσπάθησα να προσαρμοστώ και έστειλα ε, το κείμενο του ε, του πακέτου διεύρυνσης χτες το βράδυ ε, στους ευρωβουλευτές ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι ευρωβουλευτές να του ρίξουν μια ματιά αλλά πάντως σημειώνω και το θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό που είπατε και σημειώνω ότι αισθανθήκατε με αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε σήμερα. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω το πακέτο διαβρύνσης του 2010. Αλλά πριν μπω στην ουσία αυτού του πακέτου θέλω να σας παρουσιάσω κάποιες γενικές ιδέες θα σας αναφέρω κάποιες βασικές αρχές και προκλήσεις που έχω να αντιμετωπίσουμε. Θα αναφερθώ στις δύο γνωμοδοτήσεις για το Μαυροβούνιο και την Αλβανία και μετά θα παρουσιάσω τα κύρια ευρήματα από, για άλλες υποψήφιες και ενδυνάμει υποψήφιες χώρες. Ε, τούτο το πακέτο ε, ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος μιας χρονιάς στην οποία ε, συνέβησαν σημαντικά πράγματα για τις ε, χώρες διεύρυνσης δείχνει ότι κάθε χρόνο επιτυγχάνονται ε, πράγματα και κερδίζουμε πείρα που βοηθούν στη βελτίωση και την καλύτερη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διεύρυνσης οι βασικά θεμέλια και βασικές αρχές της όλης διαδικασίας παραμένουν βεβαίω η πλήρη στήριξη των κριτηρίων της Κοπενχάγης και το κονσένσο του 2006, οι δεσμεύσει που αναλαμβάνουμε και η αιρεσιμότητα που εφαρμόζεται για τις στις υποψήφιες χώρες. Α, αυτή η μεθοδολογία είναι δοκιμασμένη, έχει αποδείξει και την αξία της ε, και έφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές από τις χώρες που είναι σήμερα μέλη. Οι κανόνες του παιχνιδιού παραμένουν οι ίδιοι. Ε, αλλά βεβαίως ε, πρέπει να μάθουμε και να εφαρμόσουμε τα μαθήματα από τα αυτά που είδαμε στους τελευταίους γύρους διεύρυνσης. Ε, ξέρουμε ε, τι πώς δουλεύουν τα benchmarks για την, το άνοιγμα και το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων. Ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση, παρακολουθούμε ναι, πώς καλύπτονται, γίνονται σεβαστές κάποιες ε, αρχές και αξίες, ε, πώς γίνονται κάποιες βασικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται από τα κράτη-μέλη και ε, κάνουμε και εμείς βεβαίως την ανάλυση μας σε κάποιους κυρίους τομείς. Όταν ε, ανέλαβα τα καθήκοντά μου και ήρθα εδώ στη σχετική ακρόαση τόνισα ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να στις χώρες που είναι υποψήφιες να δίνουμε και πληροφορίες και ενημέρωση δηλαδή αλλά και συμβουλές και στήριξη και καθοδήγηση Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα χρειαζόμαστε μια διαδικασία που να υποστηρίζει, αλλά να είναι και αυστηρή και να μπορεί να θεσπίζει ελέγχους ε, που ε, θα μας δείχνουν ότι τα κριτήρια τηρήθηκαν. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και πριν να μπω τώρα κύριε Πρόεδρε στις γνωμοδοτήσεις για την Αλβανία και το Μαυροβουνίο να πω μερικά πράγματα για τη γενική έννοια της διαβρύνση και για το που εστιάζεται το έγγραφο στρατηγικής της Κομισιόν. Βεβαίω η οικονομική κρίση την οποία διατρέχουμε είναι το κύριο θέμα των ημερών ε, και μπορεί κάποιοι να αναρωτηθούν γιατί παίζει ρόλο η διεύρυνση και γιατί χρειάζεται η διεύρυνση υπό τι παρούσε συνθήκες. Είναι σημαντική η διεύρυνση, κυρίες και κύριοι, διότι ενισχύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Είναι τεράστιου στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η διεύρυνση. Και η διαδικασία διεύρυνσης μας βοηθάει να επιτύχουμε κι εμείς καλύτερα του στόχου μα σε κάποιου τομεί Βοηθάει την ανάπτυξη, την οικονομική, την βιώσιμη ανάπτυξη. Μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης. Μας βοηθάει να επιτύχουμε τους στόχους της ε, Ατζέντα 2020. Ε, Μας βοηθάει να βελτιώσουμε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τονίσουμε τη σημασία και το βάρος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο, στην Ιφίλιο. Και βεβαίως υπάρχει οικονομική κρίση, όπως είπα, και οικονομική ύφεση. Λοιπόν, η συνεργασία και ο διάλογος για οικονομικά θέματα και η στενότερη ε, οικονομική σχέση με κάποιες χώρες, αυτές τις που λέμε χώρες της διεύρυνσης, θα βοηθήσουν τα αυτά θα βοηθήσουν τα πράγματα και θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός κόσμου ο οποίος είναι ρευστός και ο οποίος έχει όχι ένα, όχι δύο, αλλά πολλαπλούς πόλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι ότι πρέπει να θεσπίσει αν δεν υπάρχει ή να κάνει στενότερη τη συνεργασία με παλιότερους ανταγωνιστές ή αντιπάλους για να μπορέσει να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του χώρου γύρω μας. Η πολιτική μας διεύρυνση ε, μας δείχνει ότι μπορούμε σημαντικές προκλήσεις να τις κάνουμε σημαντικές ευκαιρίες για να έχουμε πιο ασφαλή και ευημερούσα Ευρώπη. Πιστεύουμε πραγματικά ότι, η... ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και στη σταθερότητα, στην ειρήνη, στην καλύτερη παγκοσμιοποίηση σε μια άλλου είδους παγκοσμιοποίηση στον, κόσμο, στον κόσμο μας και για να συνεχίσουμε να είμαστε επιτυχείς θα πρέπει να, η, πολ, πολιτική μας για τη διεύρυνση να η, συνεχίσει να είναι αξιόπιστη γιατί η αξιοπιστία δεν είναι μονόδρομος είναι αμφίδρομη έννοια για τα κράτη-μέλη η αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης σημαίνει αυστηρή αιρεσιμότητα σε σχέση με τις υποψήφιες χώρες. Για τις υποψήφιες χώρες σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι 100% έτοιμες να ακολουθήσουν ορισμένους κανόνες. Θα πρέπει να μπορούν να ε, ε, δράσουν μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να αλλάξουν, να κάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και να έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα για οι συγκεκριμένες χώρες δεν θα πρέπει απλώς να κάνουν επιφανειακές αλλαγές ε, ή να αλλάζουν κάποιες νομοθετικές πράξεις ε, θα πρέπει να κάνουν πραγματικές αλλαγές να είναι 100% πρόθυμες να αλλάξουν αλλά συγχρόνως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100% πρόθυμη να συμπεριλάβει και νέες χώρες η θέση ισχύ της σύμβασης, της συνθήκης της Λισαβόνας είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για που σχετίζεται με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευρυνθεί. Ε, εάν και εφόσον αποφύγουμε ορισμένα εμπόδια που οφείλονται σε θεσμική συμφόρηση θα έλεγα τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ακολουθήσει μια διαδικασία διεύρυνσης να διατηρήσει την ορμή της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και να εξασφαλίσει ότι οι υποψήφιες χώρες που θα πρέπει όπως είπα να είναι 100% πρόθυμες να αλλάξουν να, βοηθήσουν να βοηθήσει λοιπόν αυτές οι υποψήφιες χώρες να γίνουν πλήρη μέλη οι αλλαγές που απαιτούμε από τις καινούριε χώρες είναι πολύ σημαντικές είναι αλλαγές που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, με τους θεσμούς, με τον αγώνα κατά του εγκλήματος, κατά της διαφθοράς. Ε, πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις κοινωνίες των χωρών αυτών, αλλά για τις κοινωνίες των ήδη, των χωρών που είναι ήδη κράτη-μέλη. Ε, μετά την ένταξη των χωρών, αν οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ήδη γίνει, δεν, χρειάζεται να γίνουν πολλά άλλα πράγματα. Ε, και, για, και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία οι χώρες υποψήφιε χώρες θα πρέπει να προσέξουν. Παραδείγματο χάρη ελευθερία έκφραση ε, μεσών μαζικής ενημέρωσης. Αυτά όλα τα, ε, τα πράγματα μπορεί να είναι αυτονόητα για κάποιου, αλλά δύσκολα να αλλάξουν σε κάποιες άλλες χώρες. Δημερεί ε, σχέσεις και δημερεί προβλήματα πρέπει επίσης να επιληθούν από, και από την Ένωση και από τις υποψήφιες χώρες ναι, λαμβάνοντα υπόψη τα συμφέροντα και τον μεν και των δε. Ε, επίσης η περιφερειακή συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη σταθεροποίηση και τη διαδικασία σύνδεσης. Δεν θα πρέπει να υπονομεύεται η περιφερειακή συνεργασία από διαφορές για το κοσφοπέδιο. Η απελευθέρωση του καθεστώτος χορήγησης ε, προξενικών θεωρήσεων. Ε, έχει ήδη γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος και γι' αυτό will και γι' αυτό ε, η, ήρθαν ορισμένε υποχρεώσεις για τους υπηκόους της ε, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας. Ε, χτες αποφασίστηκε ότι οι απαιτήσει για τη θεώρηση θα αρθούν επίσης και για τους κόσμους της Βοσνίας, της Ερζεγοβίνη και της Αλβανίας. Με την, ε, θα ξεκινήσει και ο σχετικός διάλογος με το Κωσυφοπαίδιο. Αλλά χρειάζονται και άλλες προσπάθειες να γίνουν. Να αναφερθώ τώρα στις γνωμοδοτήσεις για το Μαυροβούνιο και την Αλβανία. Όπω είπε κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλι υιοθέτησε τι γνωμοδοτήσεις για την Αλβανία και το Μοντενέγκρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρηση θα πρέπει να ανοίξουν με το Μαυροβούνιο και την Αλβανία Μόλι αυτέ οι χώρε έχουν επιτύχει ένα ικανοτικό επίπεδο συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξη και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή πληρούν ε, μια σειρά από προτεραιότητε κλειδιά που καθορίζονται στις γνωμοδοτήσεις. Έχουμε κάνει μια σε βάθος ανάλυση ε, αξιολογώντας κάθε χώρα ε, στη βάση ε, των δικών της στοιχείων και ισχυρών σημείων και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Η τήρηση των πολιτικών ε, κριτηρίων της Κοπεχάγης είναι αποφασιστική σημασία για το κατά πόσον θα προτείνουμε ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, ένταξης. Ενώ και οι δύο αυτές χώρες έχουν πραγματοποιήσει πρόοδο, υπάρχουν ακόμα εκρεμή ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης και πριν σκεφτούμε καν το ενδεχόμενο αυτό. Ιδιαίτερα όσον αφορά το κράτος δικαίου. Η γνωμοδότηση για το Μαυροβούνιο αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια και ε, στη θέσπιση ενός νομικού και θεσμικού πλαισίου ε, φυγραμμισμένου με τα ε, ευρωπαϊκά πρότυπα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να λειτουργεί κανονικά και να υπάρχει επικοινωνία διάλογο ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα ε, και οι σχέσεις γειτονία πρέπει να είναι καλές. Σαν αναγνώριση των ε, επιτευγμάτων της, ε, συστήνουμε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για το Μοντενέγκρο. Αυτό αντικατοπτρίζει ε, στη θέση μας ότι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί χειροπιαστά επιτεύγματα όσον αφορά την ε, πορεία προς την ε, ένταξη. Και η Αλβανία έχει πραγματοποιήσει θετικά βήματα. Ε, και η χώρα αυτή παίζει ένα θετικό ρόλο στις περιφερειακές σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, οι ε, επιτεύξεις της και θετικά σημεία ε, σε διάφορους τομείς υπονομεύονται από το πολιτικό αδιέξοδο που θέτει υποβισβήτηση τους πολιτικούς θεσμούς της χώρας. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου και έχουν μπλοκαριστεί ε, διάφορες ε, θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο για τον ε, σεβασμό των πολιτικών κριτηριών τη Κοπενχάγη. Δεν προτείνουμε λοιπόν το καθεστώ τη υποψήφια χώρα για την Αλβανία και αυτό είναι συνεπέ με την προσέγγιση μα όσον αφορά το πολιτικό διάξοδο μέχρι στιγμή. Για παραπάνω από ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και επενώ τι συνεχεί προσπάθειε που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άποψη αυτή έχει προσπαθήσει να περάσει ένα σαφές μήνυμα προς όλα τα πολιτικά κόμματα, προς όλα λέω τα πολιτικά κόμματα, είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση ε, και τα καλεί να δείξουν υπευθυνότητα και να βρουν μια λύση για το αδιάξοδο αυτό. Μια προσέγγιση λοιπόν που βασίζεται στην αξιοπιστία. Εμείς καθορίσαμε συγκεκριμένες προτεραιότητες στις γνωμοδοτήσεις παρέχοντας σε κάθε μία από αυτές τις χώρες σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, σαφή καθοδήγηση σχετικά με το τι πρέπει να γίνει. Θα αξιολογήσουμε την πρόοδο που θα έχει πραγματοποιηθεί ε, στο πακέτο του 2011 για τη διεύρυνση. Ε, θα κρίνουμε κάθε χώρα ε, ξεχωριστά, γιατί κάθε χώρα αποφασίζει την ταχύτητα με την οποία κινείται στο δρόμο αυτό προς την Ευρώπη. Θα έρθω τώρα, ε, κύριε Πρόεδρε, σε άλλε υποψήφιε και ενδυνάμει υποψήφιες χώρες. Όσον αφορά την Κροατία, οι διαπραγματεύσεις ένταξη έχουν φτάσει στην τελική φάση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την ε, πρώην Ιουγκοσλαβία ε, παραμένει μια προπόθεση για την πρόοδο της Κροατία καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτής, ε, σύμφωνα και με το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Η Κομισιόν θεωρεί ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις μόλις η Κροατία έχει ε, ε, πετύχει όλα ε, τα benchmarks, ε, τα κριτήρια που έχουν τεθεί όσον αφορά ε, το δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν αξιόπιστες επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή όλων αυτών των στοιχείων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη και μετά την προσχώρηση θα ε, ε, κάνουμε έναν απολογισμό της πρόοδου που θα έχει πραγματοποιηθεί για το σχετικό κεφάλαιο 23 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011. Η ποιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ε, διαδικασίας προσχώρησης της Κροατίας έχουν μεγάλη σημασία για ολόκληρη την περιοχή. Η Τουρκία. Η Τουρκία έχει συνεχίσει την ε, πορεία της ε, προς την ε, πολιτική μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα μέσω της μεταρρύθμισης του συντάγματός της. Χρειάζονται περαιτέρω αποτελέσματα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δημοκρατικό άνοιγμα και την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Και ιδιαίτερα η ελευθερία της έκφρασης πρέπει να εξασφαλιστεί και στην πράξη. Προχωρώντας προς την ε, εκπλήρωση των benchmarks, καθώς επίσης και ε, των προϋποθέσεων που ε, προσδιορίζονται στο διαπραγματευτικό πλαίσιο, η Τουρκία θα μπορέσει να επιταχύνει την πορεία των διαπραγματεύσεων. Είναι επίγον πλέον, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, τονίζω τον επίγοντα αυτό χαρακτήρα, η Τουρκία λοιπόν θα πρέπει επιγόντως να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για πλήρη μη διακριτική εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλου της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης. Απουσία τέτοιας πρόοδου σε αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τα μέτρα που ισχύουν από το 2006. Αυτά θα έχουν ένα ε, συνεχές αποτέλεσμα ε, πάνω στην συνολική πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, οι ηγέτες ε, της Ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής ε, κοινότητας συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για, μια, ε, για ένα συνολικό διακανονισμό του θέματος υπό την αιγίδα ε, των Ηνωμένων Εθνών. Καλό και τους δύο να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές όσο δυνατόν γρηγορότερα σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Επίσης, θα επαναλάβουμε την έκκληση μας προς την Τουρκία να συμβάλλει με συγκεκριμένους τρόπους προς ε, μια συνολική ρύθμιση του Κυπριακού. Για την Ισλανδία. Η διαδικασία ε, ένταξης της Ισλανδίας έχει ξεκινήσει. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης θα ανοίξουν τον Ιούλιο του 2010. Έχει ξεκινήσει η ανασκόπηση της νομοθεσίας της Ισλανδίας. Τα πρώτα κεφάλαια μπορεί να να ξεκινήσουν να εξετάζονται πριν από το επόμενο καλοκαίρι και η Ισλανδία θα πρέπει να αντιμετωπίσει υφιστάμενες υποχρεώσεις όπως αυτές που αναφέρονται στην ΕΦΤΑ και από την αρχή παρακολούθησης ε, όσον αφορά τον ΕΟΧ. Χρειάζονται πάρα πολλές ε, προσπάθειες ώστε οι πολίτες της Ισλανδίας να ενημερωθούν σωστά σχετικά με το τι συνεπάγεται η Ισλανδία να γίνει μέλος. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθεί να πληρεί ικανοποιητικά τα πολιτικά κριτήρια. Υπήρξε πρόοδος σε μεγάλους τομείς μεταρρύθμισης, αν και δεν είναι ε, ο ρυθμός πάντα ο ίδιος. Χρειάζονται δηλαδή μεγαλύτερες προσπάθειες για τη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Η Κομισιόν επαναλαμβάνει τη σύστασή της να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως απαιτείται ομόφωνη απόφαση από τα κράτη-μέλη για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητο να εξευρεθεί μία αμοιβαία αποδεκτή λύση για το θέμα της ονομασίας μετά από διαπραγματεύσεις. Τον Οκτώβριο του 2010 το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιό να υποβάλει την γνωμοδότησή της για τη Σερβία. Συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτική μεταρρύθμιση η Σερβία και να δημιουργήσει μια, και δημιουργεί μια πολύ καλή ε, πορεία στην εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας. Χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες στον δικαστικό τομέα και στη δημόσια διοίκηση και στην καταπολέμηση του εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Επίσης πρέπει να συνεργαστεί σε σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, διότι υπάρχουν οι δύο φυγάδες που δεν έχουν συλληφθεί. Η πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Δικαστήριο είναι διεθνής υποχρέωση. Η Σερβία πρέπει να επιδείξει μια επικοδομητική στάση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοσυφοπεδίου στο περιφερειακό εμπόριο και πρέπει να υπάρχει και συνεργασία. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τη Ιούλεξ για το κράτος δικαίου όσον αφορά το βόρειο τμήμα του Κωσυφοποντίου. Τώρα, η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη μετά τις γενικές εκλογές του Οκτωβρίου πρέπει να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις. Ειδικότερα η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη πρέπει να ευθυγραμμίσουν το σύνταγμά τους σε σχέση με το Ευρωπαϊκο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να βελτιώσει η χώρα αυτή ακόμη την αποτελεσματικότητα ε, στη λειτουργία των θεσμών της. Πρέπει δε να εφαρμόσει και τους νόμους και τους κανόνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο για την Βοσνία Ερζεγοβίνη να προχωρήσει και να υλοποιήσει τους στόχους όσον αφορά το κλείσιμο, που θα οδηγήσουν, εξελίξεις που θα οδηγήσουν στο κλείσιμο του γραφείου του ΙΠΑ του εκπροσώπου. Επίσης, χρειαζόμαστε να διευκολύνουμε το διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνας, ώστε να προωθηθεί η συνεργασία για να επιτευχθεί πρόοδος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιωθούν και οι ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι πολύ καλή ευκαιρία, όχι μόνο για διμερείς σχέσεις, αλλά για την περιφέρεια στο σύνολό της και την περιφερειακή συνεργασία. Στο Κωσυφοπαίδιο τώρα. Η διαδικασία αποκέντρωσης έχει προχωρήσει σημαντικά. Η συνεργασία με τη Γιούλεξ έχει ενταθεί, όμως μεγάλες προκλήσεις παραμένουν. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, περιλαμβάνοντας δε και τη δημόσια διοίκηση και τη δικαστική εξουσία. Περισσότερα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, το οργανωμένο κρίμα, ε, έγκλημα, με συγχωρείτε, και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Ο διάλογος και η συμφιλίωση μεταξύ των ε, κοινοτήτων και η προστασία και η ολοκλήρωση, η ολοκληρωμένη ένταξη των μειονοτήτων, ιδιαίτερα δε των Σέρβων του Κωσυφοπαδίου, ε, είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν ακόμη. Η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ανησυχητική και πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε περιφερειακές εξελίξεις. Συμπέρασμα τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, για να προχωρήσουμε στην τρέχουσα διαδικασία ολοκλήρωσης και διεύρυνσης, μας έχουμε την ευκαιρία πραγματικά να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις και πρέπει να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία και την συνέχεια αυτής της διεργασίας. Δεν πρέπει να χάσουμε την προωθητική μας δύναμη. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του 2010. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια ακόμη. Οι απόψεις που σας είπα αντανακλούν τις πεπιθήσεις της Κομισιόν, τις πεπιθήσεις προσωπικές μου και τις πεπιθήσεις πιστεύω και τις δικές σας ότι η διεύρυνση είναι ζωτική σημασίας. Προσπάθησα να διατηρήσω τις στενότερες επαφές δυνατόν μαζί σας και ελπίζω ότι αυτές οι επαφές ήταν χρήσιμες για σας και ήταν πραγματικά υποφελείς για μένα. Στην Επιτροπή σας υπάρχει τεράστια εμπειρία και μεγάλη κατανόηση όσον αφορά τη διαδικασία της διεύνησης. Κύριε Πρόεδρε, ε, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πολύ στενά προς όφελος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία, την τελευταία χρονιά έχουμε παρατηρήσει τις τεράστιες προσπάθειες των χωρών που είναι ε, να γίνουν μέλη. Αλλά Υπάρχουν μεγάλη πρόοδος, αλλά υπάρχουν και κρεμότητες. Χρειάζονται όμως οι χώρες αυτές την υποστήριξή μας. Έχουν τη δικιά μας και είμαι σίγουρος ότι θα έχουν και τη δικιά σας υποστήριξη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο ομιλητών για να εξοικονομήσουμε χρόνο και να δώσουμε προτεραιότητα στα πιο λεπτά ζητήματα, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να δώσουμε κατά πρώτο λόγο του, το λόγο στους συζητητές που ετοιμάζουν τις εκθέσεις για τις διάφορες χώρες και στη συνέχεια στους συντονιστές. Ε, ε Έλμαν Ρόιτεν λοιπόν ο, ο, και ο κύριος Σαλαφράγκα. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ, ε, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά που ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί και να κάνουμε κατάχρηση του χρόνου που μας ε, αφιερώνει ο, ο κύριος Επίτροπος. Νομίζω ότι έχετε αποδείξει την καλή σας ε, θέληση απέναντι στην Επιτροπή μας και είναι προφανές ότι είστε ανοιχτός στην επικοινωνία. και θα ήθελα να πω ότι ίσως ε, τα, οι άλλοι επιτροποί δεν κάνουν ε, το ίδιο, δεν ακριβούν, δεν ε, ακολουθούν ακριβώς το παράδειγμά σας. Ε, θα σας κάνουμε λοιπόν όλες αυτές τις ερωτήσεις, ίσως κάνοντας μια κάποια κατάχρηση του χρόνου σας. Πριν από πέντε χρόνια οι σχέσεις μας με την Τουρκία βρίσκονταν εν εξελίξη και Υπήρχαν κάποια καλά σημεία και κάποια πιο σκοτεινά. Ε, ζητήσαμε θεσμικές ε, ε, βελτιώσεις, βελτιώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις όσον αφορά την ισορροπία ανάμεσα στην στρατιωτική και την πολιτική εξουσία. Ε, Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν ε, κάποια άλλα σημεία που παρέμειναν σκοτεινά και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο καμπής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν σε ποιο βαθμό για να ξεπεράσουμε ας πούμε Είπα ότι βρισκόμαστε σε σημείο καμπής και σε, όχι, όχι σε αδιάξοδο, αλλά μέσα σε πέντε χρόνια διαπραγματεύσεων τρία κεφάλαια άνοιξαν και φαίνεται ότι είναι αδύνατο να ανοίξουν άλλα κεφάλαια. Ε, και όσον αφορά την εξομάλυση των σχέσεων με την Κύπρο, σε ποιο βαθμό ε, παίζει το θέμα αυτό ε, κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις συνθήκες δεν θέλω να αφιζητήσω τα θετικά βήματα της Τουρκίας μέχρι τώρα. Σε ποιο βαθμό το ζήτημα αυτό, το κυπριακό δηλαδή, ε, σκιάζει την όλη διαδικασία. Δεύτερον, στις διαδικασίες ε, με την Τουρκία, ε, πώς, ε, ε, τι έχουμε να πούμε για το θέμα της συμφιλίωσης με την Αρμενία. είχαμε κάποια βήματα πέρυσι, έγινε μια επικύρωση των πρωτοκόλων που απαιτούνται για να προχωρήσει περαιτέρω αυτή η υπόθεση. Σε ποιο βαθμό επίση, οι σχέσεις τη Τουρκία με το Ιράν ε, είναι πηγή ανησυχιών. Και ε, σε ποιο βαθμό ε, δυσκολεύονται οι διαπραγματεύσεις μας λόγω αυτών των εξέλιξεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάποντα που είναι εισηγητής για την Κροατία. Για δυόμιση λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, κύριε Πέτροπε, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε εκ των προτέρων, Πολύ σημαντικό αυτό. Σε γενικέ γραμμέ η έκθεση είναι πολύ ισορροπημένη και αναφέρεται στα κυριότερα προβλήματα. Για την Κροατία τονίσατε το πρόκειται για το ελληνικό στάδιο. Υπάρχουν ορισμένε επικρίσει ε, στην Κροατία αυτή τη στιγμή και πριν από την ε, συνέψη τύπου, ότι δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη ημερομηνία. Από την άλλη μεριά είναι σαφέ νομίζω ότι το θέλουμε να γίνει το γλυγορότερο δυνατόν. Είναι σαφέ ότι θα είναι καλό να έχουμε την ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων στο πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτου, Από εκεί και πέρα όμω η Κροατία είναι εκείνη που θα πρέπει να καταβάλει τι περισσότερε προσπάθειες. Για δύο θέματα που αναφέρατε, όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση δικαιοσύνης ε, του δικαστικού συστήματος, ε, το θέμα της καταπλώμησης διαφοράς. Αυτά είναι θέματα για τα οποία πρέπει να τους πούμε κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε και μετά θα συμφωνήσουμε. Θεωρητικά είναι αδύνατο να κάνουμε ίσως οτιδήποτε άλλο. Η Κροατία πρέπει όμως τώρα να δράσει όσον αφορά τον πολιτική ανταγωνισμού, ιδίως για τα ναυπηγεία και εκεί πρέπει κάτι να κάνουμε. Αλλά φαντάζομαι ότι αναγνωρίζουμε ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε όπως θα θέλαμε. Αλλά όπως σας είπα και αυτό είναι δικό του θέμα. Συμφωνώ λοιπόν με την έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής και το μήνυμά μου προς την Κροατία είναι πάρε τα όλα σοβαρά, κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε και τότε θα μπορέσουμε ίσως να ολοκληρώσουμε το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλερ, ο οποίος είναι η δυόμιση λεπτά. Grazie, ε, Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar File, za... Σας ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για την έκθεσή του, για την εργασία του. Γιατί η παρουσία σας κατέδειξε τι ε, πραγματοποιήσατε το περασμένο έτος και θέλω να υποστηρίξω τις προσπάθειές σας όσον αφορά τη συνεργασία με τη, τα κοινοβούλια. Είναι σωστό να μιλάει με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση τι υποψήφιε χώρε και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα πρέπει δηλαδή να συμφωνούν. Όσον αφορά τη Μακεδονία, η Κομισιόν θεωρεί ότι η Μακεδονία πληρεί τις πολιτικές προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να προχωρήσει όσον αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ, το δικαστικό και θα πρέπει η Κομισιό να παρατηρήσει προσεκτικά το θέμα της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τομέα αυτός για την δημοκρατία στις χώρες αυτές. Ε, πέρσι, από ό,τι θυμάμαι, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Είχαμε μιλήσει για ένα παράθυρο ευκαιρία. Είχαμε πει ότι είναι θέμα μόνο χρόνου ότι θα μπορούσε μετά από πέντε χρόνια να ξεκινήσει διαπραγματεύσει στη Μακεδονία. Τώρα η αισιοδοξία αυτή εξαφανίζεται. Από ό,τι φαίνεται βρισκόταν στη σωστή άγουστα η Μακεδονία, αλλά με την ε, διαμάχη της, με την Ελλάδα, λόγω του ονόματος δηλαδή, παρεμποδίστηκε η πρόοδος και θα πρέπει να έχουμε το γλυγορότερο δυνατόν τη λύση, αυτή είναι η σύσταση, αλλιώς αδίκως η Μακεδονία θα παραμείνει πίσω. Θέλουμε ένα συμβιβασμό με περισσότερη ευελιξία και από μακεδονικής και από ελληνικής πλευράς. Θα ήθελα ιδίω να υποστηρίξω αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει πραγματικά να ληφθεί υπόψη αυτό το σημείο. Γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα συμφέροντα της Ελλάδας και τα συμφέροντα της Μακεδονίας και θα πρέπει η Κάθριν Εστων, η υπατή εκπρόσωπος και εσείς ως επίτροπος να προσπαθήσετε από κοινού να καταβάλλεται περισσότερες προσπάθειες και προς τις δύο πλευρές για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα περισσότερο. Ίσως θα μπορούσαμε να ε, έχουμε κατά νου κάποια διαιτησία. Ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να προσφέρει συμπληρωματικές υπηρεσίες και να μην περιμένει δηλαδή διαιτησία από τα Ηνωμένα Έθνη. Και ελπίζω από κοινού να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το να γίνει η Μακεδονία κράτος μέλος. Ευχαριστώ. Βουλευτής Ρέντε που είναι ε, εισηγητής για την Ισλανδία. Σας ευχαριστώ πρώτα. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο που μου έχει χορηγηθεί. Ένα πράγμα θα πω. Καταρχήν θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την Άνοιξη αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει την απλουστευμένη διαδικασία για να μπορέσει η Ισλανδία να ωφεληθεί το γλυγόρο των δυνατών από το μέσο της ε, προεταξιακής στήριξης. Αυτό ήταν μια ομόφωνη ψηφοφορία και θα έκανε ό,τι μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διατεθούν οι πόροι αυτοί προς την Ισλανδία πριν από μερικές μέρες όμως, ανακάλυψα ότι πολλοί από τους υπουργού της κυβέρνησης που ζήτησαν να ανοίξουν διαπραγματεύσεις και που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή, ε, θεωρούν ότι τα χρήματα από αυτό το ο, προενταξιακό μέσο είναι μόνο προπαγάνδα. Και πολλοί ε, στην Ισλανδία θεωρούν ότι η χρήση αυτού του μέσου είναι επικίνδυνη για την Ισλανδική κοινωνία. Έχουμε μια καλή περιγραφή πολιτική, δηλαδή από την μεριά είναι ανοιχτή η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση, θέλει την Ένωση, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια καχυποψία όσον αφορά τη διάδοση πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς κύριε Επίτροπε, πώς ε, εξετάζετε αυτό το τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Γιατί δεν έχουμε μόνο μια πολιτική τάξη, μια κυβέρνηση που λέει ναι για την ε, διαδικασία ένταξης. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως και η κοινωνία, οι πολίτες που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι αυτή η ένταξη και τι είναι αυτό το μέσο το προενταξιακό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώντα την κυρία Πακ, που είναι εισηγήτρια για τη Βοσνία Ζεγοβίνη, θα πάρει το λόγο ο κύριος Μπρόκ για δυόμιση λεπτά. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να αντικαταστήσω την κυρία Πακ στη ζωή μου. <laughs> Τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω να το τολμήσω το εγχείρημα αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Η εξέλιξη στα Βαλκάνια εξαρτάται βέβαια πάρα πολύ σε όλες τις χώρες όσον αφορά την προοπτική ένταξη τους και για την Κροατία και ε, για την ε, ε, Βοσνία θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούν να προχωρήσουν πολλές φορές μπορεί να υπερβάλλει κανένας Πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά για τη Βοσνία. Για τη Βοσνία και τη Ροζεγοβίνη γενικά θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς το ψήφισμά μας του Ιουνίου 2010 και Απριλίου 2009 δεν οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στα κεντρικά θέματα. Δεν μπορεί να λυθεί το θέμα ούτε από τις υπηρεσίες της ΥΠΑ της εκπροσώπου πρέπει βέβαια να μην ξεχνάμε ότι λόγω τη σύνθεση τη χώρα αυτέ με τι τρει εθνικέ ομάδε και την, όλη τη δομή τη χώρα. αυτή η χώρα έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα, ιδίω στο συνταγματικό τομέα, αλλά και όσον αφορά την ε, αστυνομική συνεργασία και άλλου τομεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε όσον αφορά το θέμα των θεωρήσεων των διαβατηρίων. Και έτσι να αποστείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν έχουμε ξεχάσει τη χώρα αυτή και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ούτε ώστε θεωρώ ότι ψυχολογικά είναι πάρα πολύ σημαντικό που η Βοσνία Χαζεγοβίνη και η ε, Αλβανία μπαίνουν σε αυτόν τον κατάλογο των χωρών ε, που δεν χρειάζονται θεώρηση για τις χώρες Έγγεν. Αν λέτε ότι τονίζεται περισσότερο από τις ε, παλαιότερες διευρύνσεις το θέμα της διαφθοράς, το θέμα της δημόσιας διοίκησης, το θέμα της ε, περιφερειακής συνεργασίας, έτσι είπατε σε εισαγωγικά. Αυτά ισχύουν ιδιαίτερα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και θα ήταν καλό να υπάρχουν ορισμένα benchmarks ε, στον μισό αυτός, ιδίως όταν εξετάζουμε το θέμα της εταιρικής σχέσης. Και, εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω, θα πρέπει να σκεφτείτε κάποια στιγμή πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να παραμείνει μια χώρα όμοιρος της ε, αντιπολίτευσης στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπρόκ. Ο κύριος Κάτσινγκ, εισηγητής για την Σερβία, ε, για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. želim pozdraviti jasen jezik, ki Πρόεδρε, αγαπητέ επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που πετύχαμε μέχρι στιγμή είναι να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Η... ζητήθηκε η άποψη Τη Κομισιόν και το Βελιγράδι έχει την δυνατότητα να σκεφτεί τα θέματα της πολιτικής. Δεν είναι ποτέ μια πρόκληση υπερβολική εάν ο στόχος είναι μια θετική αξιολόγηση από την Κομισιόν. Το πρόβλημα με, την, με το κοσυφοπαίδιο μας κάνει να καταλάβουμε ότι το κύριο θέμα είναι το δικαστικό. Θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης και θα πρέπει να ξανεκταστεί όλο το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Θα πρέπει επίση να προωθήσουμε την ανεξαρτησία και την ελευθερία των ΜΜΕ. Εκεί υπάρχουν μεγάλα εμπόδια. Μονοπόλιο της ιδιοκτησίας, το θέμα τη ε, ηγεσία ε, των κομμάτων, ε, ο κίτρινο τύπο, Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πολιτική και για περαιτέρω επιβολή της δημοκρατικής κουλτούρας φιλελεύθερος θα πρέπει να αναφερθώ στο θέμα της προστασίας των ατόμων. Γιατί δεν έχει υιοθετηθεί σχετική νομοθεσία σύμφωνα με τα πρότυπα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους πολίτες του Μαυροβονίου όσον αφορά την θετική εκτίμηση της Κομισιόν για την αίτησή τους ε, ε, ένταξης. Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλες τις γειτονικές χώρες του Μαυροβονίου που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το Μαυροβούνιο θα μπορεί να είναι και ένα πρότυπο για το πώς πραγματοποιεί τις μεταρρυθμίσεις μια χώρα. Τρεις ε, γείτονε Σερβίας είναι ήδη υποψήφιες χώρες. Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μετά την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίων για την Βοσνία Ζεχοβίνη και Αλβανία θα πρέπει να δώσουμε την ίδια δυνατότητα και στην Τουρκία. Και δύο λόγια για τη Μακεδονία. Υπάρχει ακόμα το πρόβλημα του ονόματος της χώρας αυτής και θα ήθελα να καλέσω την πολιτική ηγεσία της Μακεδονίας να μην κάνει τίποτα που θα διακυβεύσει τον συμβιβασμό. Γιατί πρέπει να υπάρχει συμβασμό για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει ένταξη. Τάνεκ, εισηγητή για το Μοντενέγκρο. Θα μιλήσω και σαν συντονιστή της ομάδας μου και εκ μέρους του εισηγητή για το Μοντενέγκρο. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρώτη σας έκθεση για τη διεύρυνση και για τις γνωμοδετήσεις σας για την Αλβανία και την Μοντενέγκρο και ελπίζουμε ότι και η Κροατία θα μπορέσει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια. Αν είναι δυνατόν και η Ισλανδία αν ο λαός συμφωνήσει με δημοψήφισμα και αν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της αλίας της φάλαινας που είναι διμερές ε, πρόβλημα το Ηνωμένο Βασίλειο. Χαίρομαι για το σχόλιο σας για την Μακεδονία και παρατρύνω την Ελλάδα να βρουν μία λύση και ένα συμβιβασμό για αυτό το ακατανόητο θέμα, τουλάχιστον για φιλέλληνες σαν και μένα επαναλαμβάνω και εγώ τη σύστασή σας προς την Τουρκία, δηλαδή να ε, επηρεάσει τις συζητήσεις της ειρηνευτικής στην ε, Κύπρο, ώστε να λυθεί το, η τραγωδία αυτής της χώρας νησιού. Για το Μοντενέγκρο είναι μια μικρή χώρα, είναι θετική η γνώμη σας και είναι βεβαίως πολύ εύκολο να βρούμε ε, θετικές πτυχές, αλλά πρέπει να πω ότι εργάζεται ε, εντατικά για να προχωρήσει τις φιλοδοξίες της για το ΝΑΤΟ. Δεν συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα να μην ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν τα κεφάλαια τα οποία ζητούν τη μεταγραφή κανόνων σε εθνικό δίκαιο και κλείνουν όταν αρχίζει η εφαρμογή. Εν πάση περιπτώσει, εσείς έτσι εφαρμόζετε τη συνθήκη σήμερα ή τσερμινεύετε μάλλον και έχουμε ένα πρόσθετο εμπόδιο για το Μαυροβούνιο όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης. Εάν οι προθεσμίες είναι μικρές, 12 με 18 μήνες, ε, οι συστάσεις αυτές είναι βιώσιμες προς το Συμβούλιο. Σε γενικά υποστηρίζω θετικά τις απόψεις σας, αλλά θα ήθελα το Μοντενέγκρο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, όχι ε, πολύ αργότερα. Ευχαριστώ, Κόντι, ε, δυόμιση λεπτά, για την Αλβανία. Χουντής, με συγχωρείτε. Και η έκθεση του Επιτρόπου για τα ζητήματα της διεύρυνσης ήταν αρκετά αναλυτική, διεξοδική και πραγματική. Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Επίτροπε, Υπάρχει ένα ερώτημα που διαπερνάει τις περιπτώσεις όχι μόνο της Αλβανίας, αλλά και άλλων χωρών. Και το ερώτημα είναι το εξή. Για την Αλβανία πράγματι το πολιτικό αδιέξοδο έχει μπλοκάρει τις μεταρρυθμίσεις και αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα. Για τη Φύρο υπάρχει το θέμα της ονομασίας. Δυστυχώς και ο πρόεδρος της Επιτροπής και αρκετοί συνάδελφοι το έχουν λύσει θεωρώντας ότι έτσι πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Για άλλες χώρες υπάρχουν άλλα θέματα. Και το ερώτημα είναι, η πολιτική της διεύρυνσης που ακολουθεί, όχι επί της θητείας σας μόνο κύριε Φούλε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι αποτελεσματική, γιατί δεν είναι ελκτική σε ορισμένες χώρες να λύσουν κάποια προβλήματα που πραγματικά, αν δεν λυθούν, δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Τουρκίας που συνεχίζει να μην σέβεται, να μην τηρεί τις υποχρεώσεις και όμως συνεχίζεται μια συζήτηση και δεν γίνεται αξιόπιστη θα έλεγα πίεση ή δεν είναι ελκτική ή δεν αποτελεί κίνητρο ενδεχομένως για κάποιες χώρες το να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνοντας τα αντίστοιχα μέτρα. Θα έλεγα ότι ίσως ορισμένες φορές η πίεση δεν ασκείται προς την σωστή κατεύθυνση και βεβαίως είναι θέμα της κάθε χώρας πώς θα αντιδράσει. Επανέρχομαι στο επίδικο θέμα περί της ονομασίας της Φύρο. Δεν κατάλαβα τώρα προς τα πού πρέπει να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ελληνική πλευρά που το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων έχει μετατοπίσει τη θέση του από παλιότερη αδιάλεκτη θα λέει κανείς θέση και έχει κάνει μια συμβιβαστική πρόταση ή προς την κυβέρνηση της Φύρο. Προς τα πού θα πιέσετε για να λυθεί το πρόβλημα για να μπορέσουν να ανοίξουν οι δρόμοι. Στην περίπτωση της Τουρκίας τι συζητάτε ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες τι συζητάτε. Θα δοθούν διάφορα ή άλλα ανταλλάγματα στην περίπτωση που η Τουρκία δεχτεί να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Αυτό λοιπόν το ερώτημα, το βασικό ερώτημα με απασχολεί, ξέρω ότι σας απασχολεί και εσάς και το συνοψίζω για άλλη μια φορά. Μήπως δεν είναι αξιόπιστη η πολιτική της διεύρυνσης ούτω ώστε πράγματι τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια που τίθενται και τα αναφέρατε και δεν έχω καμία αντίρρηση οι χώρες νομίζουν ότι μπορούν να τα διαπραγματευτούν ε, κατά το δικό τους τρόπο και όχι να τα εφαρμόσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Λούνατς, εισηγήτρια για το δυόμιση Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω και σαν συντονίστρια των πρασίνων για τις ε, εξωτερικές υποθέσεις αλλά και για το Κωσυφό Πέδιο. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα για το θαυμάσιο πλαίσιο που δημιουργήσατε όχι μόνο με τη δικιά μου την πολιτική ομάδα αλλά με όλες τις πολιτικές ομάδες και τους ευρωβουλευτές. Είναι πραγματικά μια θαυμάσια βάση για τον κοινό μας στόχο τη προώθηση της διεύθυνσης. Θα ήθελα ακόμη να σας ευχαριστήσω για τη σαφήνειά σας στο λόγο. Ε, είναι τα μηνύματα σωστά αλλά και πολιτικά ε, θέλουμε να προωθήσουμε τη διεύρυνση και να καταπολεμήσουμε την κόποση σε σχέση με τη διεύρυνση που διαπιστώνουμε σε ορισμένες χώρες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά και χαίρομαι για τη φράση σας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την κινητήριά μας δύναμη να μας εγκαταλείψει. Μια ερώτηση έχω για σας. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι 100% έτοιμη πριν από τη διεύρυνση. Τι σημαίνει αυτό, τι εννοείται δηλαδή, γιατί με τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν τα καταφέραμε όλα όσα θέλαμε. Και, θέλαμε να είμαστε έτοιμοι, χρειαζόμαστε πολιτική ένωση πιο στεναρή κτλ. Δεν θέλω να περιμένω, δεν θέλω να περιμένω ας πούμε όλες τις μεταρρυθμίσεις να γίνουν προτού ενταχθούν άλλες χώρες, Ισλανδία ή δεν ξέρω ποιε άλλε. Σας παρακαλώ να αποσαφηνίζετε. Είπατε επίσης ότι ένα κλικ δεν φτάνει για να βεβαιώσουμε την εφαρμογή μέτρων. Επικρίνεται θέματα που αφορούν την ελευθερία του τύπου, την ισότητα των φίλων, τη διαφθορά κτλ. Υπάρχουν πολλά θέματα που είναι θέματα κεκτημένα και πρέπει να υλοποιηθούν και σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας. Για το κοσυφοπέδιο τώρα. Κάνατε καλή δουλειά, περιγράψατε την κατάσταση, την πρόοδο που έχει υπάρξει, την καλή συνεργασία με τη Γιούλεξ. Θα έλεγα ότι σας παρακαλώ όταν μιλάτε με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να πείτε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους δικαστές στη Γιούλεξ από τα κράτη-μέλη. Δεν έχουν αρκετούς δικαστές. Αν πρόκειται να ε, λειτουργήσει σωστά η Γιούλεξ θα πρέπει τα κράτη-μέλη να στέλνουν τους δικαστές. Είναι το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Περιλαμβάνει το κοσυφοπαίδιο. Χαίρομαι που οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν με το κοσυφοπαίδιο ε, η Σερβία έχει λάβει το μήνυμα, χρειάζεται μήνυμα και για το κοσυφοπέδιο και οι νέοι του κοσυφοπεδίου προσανατολίζονται προς την Ευρώπη, δεν πρέπει να μείνουν πίσω. Σας ευχαριστώ επίσης που ζητήσατε από τη Σερβία να είναι επικοδομητική στη στάση της προς το κοσυφοπέδιο. Κύριος Κούκαν, πρόεδρος της Επιτροπής για τις σχέσεις με τις χώρες ε, της Νότιας Ευρώπης. Πρέπει να περικόψω το χρόνο σας στο 1,5 λεπτό. Μια στιγμή. Κάποιος ζητάει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να πω. Καλύτερα να στείλετε την Επιτροπή στο σπίτι της και να έχετε τη συνεδρίαση μόνο με τους ισοεισηγητές. Πιο εύκολο θα ήταν αυτό. Κύριος Κούκαν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η εικόνα που παρουσιάσετε για τη διεύρυνση νομίζω ότι ήταν πολύ ρεαλιστική και πολύ ακριβής. Πολιτικά νομίζω ότι ήταν πολύ προσγειωμένη η προσέγγιση και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Για να αποδείξω ακόμα και τώρα ε, μετά την επιστροφή μου από τα Τύρανα ότι τα συμπεράσματά σας για την Αλβανία ήταν σωστά είδαμε ε, ότι στον διαπολιτικό διάλογο επιτέχθη πραγματική πρόοδος. Αλλά όσον αφορά το, την πολιτική κρίση, το πολιτικό διέξοδο, το εμπόδιο που υπάρχει εδώ και τόσο καιρό, είναι εντελώ παγωμένη η κατάσταση χωρίς την παραμικρή ένδειξη ότι πρόκειται να επιληθεί αυτό το πρόβλημα σύντομα. Το συμπέρασμά σα, λοιπόν για την Αλβανία είναι πραγματικά ακριβές. Η κατάσταση στα Βαλκάνια είναι τέτοια που δίνει κάποιες ευκαιρίες για τις χώρες αυτές να δείξουν πόσο σοβαρές είναι ε, όσον αφορά την ενίσχυση, το ρόλο του στην ενίσχυση της περιφερειακής ε, ε, συνεργασίας. Θα γίνουν εκλογές στο Κωσυφοπαίδιο. Η Σερβία θα έπρεπε να συμβαλεί επικοδομητικά στη διαδικασία αυτών των εκλογών. Ο διάλογος ανάμεσα στη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο θα πρέπει να αρχίσει. Η Αλβανία θα πρέπει, θα πρέπει να υποφεληθεί από αυτή την ευκαιρία για να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο αν δεν το κάνουν αυτό μόνοι τους, ίσως θα μπορούσαμε πολύ απαλά και ήπια να τους ε, πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Ο κύριος Φλούτρεν, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για 1,5 λεπτό. Παραλίγο να με πείτε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο Μιλτής. Η κυρία. Λοιπόν, στην έκθεση ε, ε, της Κομισιόν για την Τουρκία υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία σχολιάζονται εδώ και μέρες ήδη από τον τουρκικό τύπο και αφορούν πολύ καυτά θέματα ε, το μέλλον του νέου συντάγματος, η απαραίτητη συνένεση, το δημοκρατικό άνοιγμα, το κουρδικό, το εργόνεκον υπάρχουν ε, ε, πάρα πολλά θέματα που μπορούν πραγματικά να εμπλουτίσουν τη συζήτηση που γίνεται στην Τουρκία και πολλοί εμπλέκονται στη συζήτηση. Αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το, τα σχόλιά σας και προηγουμένως και αυτά που είπατε εδώ ε, σχετικά με την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάποια στοιχεία που δεν είναι και τόσο καινούρια. Είπατε ότι υπάρχουν βήματα πρόοδου, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη και είπατε ότι πρέπει να εφαρμόσει η Τουρκία το πρόσθετο πρωτόκολλο. Όλα αυτά δεν είναι καινούρια. Με την εξαίρεση μιας λέξης που ξαφνικά εμφανίζεται ε, λέτε ότι είναι επίγον πλέον το θέμα. Πιέζετε, πιέζετε και λέτε ότι η κατάσταση είναι επίγουσα. Από τι αποτελείται αυτή η επίγουσα κατάσταση. Η ανυπομονησία σας πλέον, το άγχο σας να προχωρήσουν διακασίες ε, διαπραγμάτευσης. Τι είναι αυτή, η, αυτό το επίγον. Η, βασίζεται στην ανακοίνωση των ε, Ηνωμένων Εθνών ε, που λέει ότι κουράστηκαν πλέον να περιμένουν. Η ανυπομονησία σας οφείλεται στο γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υιοθέτησε ακόμα την σύστασή σα για το άνοιγμα του εμπορίου με την Κύπρο. Και αν ε, ο ΙΕ δεν καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα στην Κύπρο, έχετε ένα σχέδιο Β, όπω το λέει πλέον ο τύπος, διότι είναι κοινό μυστικό πλέον. Ε, ο, ο τύπος μιλάει για μυστικές διαπραγματεύσεις, δεν πρόκειται για μυστικό. Ο κύριος Βίγγενεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαν σοσιαλιστές εμείς κατανάμουμε ε, δίκαια το έργο μας και είμαστε και πειθαρχημένοι. Δεν συμμετέχω ούτε σαν ομιλητής ούτε σαν συντονιστής αντικαθιστώντας κάποιον εισηγητή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Κύριε Φίλε, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών, σας χαιρετίζω για το έγγραφο που μας προτείνετε, για τις εκθέσεις σας, καθώς επίσης και για τη δουλειά που παρέχετε περίπου ένα χρόνο για τη διεύρυνση. Ως Επίτροπος για τη διεύρυνση νομίζω ότι έχετε ε, προσθέσει αλληλεγγύη και κατανόηση σε αυτή την πολιτική. Συμφωνούμε ότι η διεύρυνση δεν είναι μόνο μια διοικητική λειτουργία πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι μεταδίδουμε σημαντικά πολιτικά μηνύματα που ενθαρρύνουν περιοχές. Στη χρονιά που μας πέρασε το πράξατε αυτό. Η φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων είναι καλό και εκτιμένο. Η απόφαση για τη Σερβία και το Μοντενέγκρο δίνει περαιτέρω βεβαιότητα στα κράτη ότι δεν σταματάει αυτή η διαδικασία, συνεχίζεται και εάν τα κράτη ακολουθήσουν δίκαια πολιτική θα τα καταφέρουν. Όμως η διεύρυνση πρέπει να έχει και υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Ε, έχετε κατά νου πρόσθετα μέτρα για να ενημερώσετε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρησιμότητα της διεύρυνσης. Πολύ σωστά υπογραμμίζετε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη της ε, κοινωνικής ολοκλήρωσης σε σύντομο μέλλον προβλέπετε συμπληρωματικά μέτρα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριο Λάμστροφ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα να πω για τις εισαγωγικέ σα παρατηρήσει ότι μου φαίνεται ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της διαδικασίας ε, ε και το καλωσορίζω αυτό. Έχει πληγεί η εικόνα ε, λόγω της, ε, της ερεσιμότητας, της απορροφή τι τις δυνατότητες απορρόφησης των κονδυλίων ε, κλπ. Ε, είχαμε ε, το 2004 μια διάβρεση και δύο χώρες προσχώρησαν ανεξάρτητα από το βαθμό προετοιμασίας που είχαν επιτύχει. Χρειάζεται λοιπόν να αποκαταθεί η αξιοπιστία της ε, και ευχαριστούμε για, που υποστήριζε αυτή τη θέση. Ε, η, Επισημένω ότι δεν αναφέρεται καμία ημερομηνία για την Κροατία. Κάποιοι συνάδελφοι διαφωνούν, αλλά εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προσέγγιση. Για την Τουρκία διάβασα την έκθεση. Επιλέξατε πολύ προσεκτικά τα λόγια σας, αλλά δεν τα μασίσατε. Και το καλωσορίζω και αυτό. Η συνάδελφος ρωτάει πού είναι ο επίγον χαρακτήρας όταν υπάρχουν μόνο τρία κεφάλαια που απομένουν. Ε, πολύ σωστή λοιπόν είναι αυτή η ερώτηση. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε αυτή την προσέγγιση. Ήταν μια πολύ καλή αρχή αυτή σήμερα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό για τον κύριο Χατζηγεωργίου. Να σας καλωσορίσω και εγώ κύριε φίλε στην Επιτροπή μας. Θα πω εξ αρχής ότι οι ερωτήσεις που είχα στο μυαλό μου και που αφορούσαν την Τουρκία έχουν ήδη ελεχθεί από συναδέλφους. Ε, κυρίως οι ερωτήσεις που έχουν το τοποθετηθεί από τον κύριο Σαλαφράγκα. Ο λόγος που θα επανέλθω είναι γιατί θέλω πάρα πολύ ειλικρινά να σας ενθαρρύνω στο να χρησιμοποιήσετε όσα όπλα έχει στη διάθεση του το γραφείο σας όπως ακριβώς είχατε πει στην πρώτη μας συνάντηση εδώ για να επιληθεί το Κυπριακό και να μπει η Τουρκία σε πορεία ένταξης. Υπάρχουν στον αέρα πληροφορίες για μυστικές διαβουλεύσεις. Θέλω μόνο σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα να σας υποδείξω, να σας πω μην βάλετε στο τραπέζι την ιδέα του ανοίγματο παράνομα κατεχόμενου εδάφους της Κύπρου ως αεροδρόμιο για την τουρκοκυπριακή κοινότητα γιατί θα καταρρεύσει οποιαδήποτε σκέψη ή προσπάθεια έχετε στο μυαλό σας για να κινηθούν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχετε όμως όπλα και θέλω να σας πω ότι η Κύπρος και η κυβέρνηση και τα κόμματα υποστηρίζομαι και είμαστε ειλικρινείς. Ονορεύωρε Γιαννάκου un Κυρία Γιαννάκου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον Επίτροπο ε, και τον συγχαίρω για τις εκθέσεις του, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικές. Το ερώτημα που παραμένει βέβαια είναι ε, ότι οι χώρες αυτές λίγος πολύ έχουν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία με την ένταξή τους κάποια στιγμή θα μεταφερθούν μέσα στην Ένωση. Είπατε κύριε Επίτροπε ότι δεν μπορούμε συνεχώς να θέτουμε αυτά τα προβλήματα μπροστά. Πρέπει ε, κατά κάποιο τρόπο να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Όμως αυτά δεν χάνονται, θα παρουσιαστούν. Παραδείγματος χάρη υπόθεση του Κόσοβο δεν μπορεί ε, να μην είναι πρόβλημα αποκλείεται να λυθεί απλώς με συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Και το ίδιο δεν μπορεί να λυθεί η κατάσταση στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου η συμφωνία του Ντέιτον φαίνεται σε όλο το μεγαλείο ότι απέτυχε. Αυτά τα προβλήματα πώς αντιμετωπίζονται. Onorevole Severino, un minuto. Ο κύριος Σεβερίν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το έγγραφο αυτό και πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να έχουμε μια στρατηγική ε, οπτική. Ο μόνος τρόπος για να έχει όραμα και αξιοπιστία η διαδικασία αυτή. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι θα έπρεπε στο έγγραφό σας να περιλάβετε μια αξιολόγηση και του παρελθόντος και των διδαγμάτων του παρελθόντος. Ένα από αυτά τα διδάγματα είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε στην άκρη τους ανθρώπους, τις κοινωνίες, τους λαούς. Μόνο τα τεχνικά ε, ε, ζητήματα δεν είναι αρκετά για να βελτιωθεί ε, η κατάσταση του λαού. Δεύτερον, δεν πρέπει να αφήσουμε τα προβλήματα στα κράτη-μέλη. Γιατί οι ε, του παρελθόντος ε, δεν ήταν αποτυχία, ήταν μια επιτυχία. Αλλά σαν αποτυχία πολλές φορές γίνονται αντιληπτές μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν τα ίδια τα κράτη να προετοιμάζονται. Και πρέπει πιστεύω να προσδιορίζουμε γιατί η διεύρυνση είναι μια ανάγκη και για μας και όχι μια ανάγκη μόνο για τις υποψήφιες χώρες. Και τέλος, θα πρέπει να ε, περιλάβετε και κάποια ε, διορθωτικά μέτρα με τα ενταξιακά για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της όλης διαδικασίας. Watson, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι αν μπορώ να ρωτήσω ε, ειδικά τον Επίτροπο για την Τουρκία και για την Κύπρο. Ο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σας συμβουλεύτηκε, κύριε Επίτροπο, προτού καλέσει τον κύριο Χριστόφια και τον κύριο Έρογλου στη Νέα Υόρκη και σε ποιο στάδιο η Βόρεια Κύπρος γίνεται υπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για τον ΟΗΕ. Ο κύριος Πόσελτ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, καταρχήν όσον αφορά την Κροατία, το κοινοβούλιο είναι αντιθέσει προς τον συνάδελφο Κλάμψοφ ζήτησε οι να ολοκληρωθούν το αργότερο το επόμενο έτος. Και χωρίς να αναφέρεται η ημερομηνία, θα ήθελα να σα ρωτήσω, θεωρείτε ότι θεωρητικά αυτό είναι δυνατό, ότι η Γκρική Προεδρία του Συμβουλίου θα μπορέσει να ολοκληρώσει αυτές τις διαπραγματεύσει. Εγώ πριν από εβδομάδα ήμουν στον τρέο συνάδελφό μα ε, Σμιτ, ε, που είναι τώρα πρόεδρος του, του Συμβουλίου, που είναι αποφασισμένος να το κάνει, αλλά δεν ξέρω αν το θεωρείται δυνατό. Μετά, για την Μακεδονία, ε, θυμίζουμε στην Ελλάδα την προσωρινή συμφωνία που είχε αναλάβει την υποχρέωση διμερεί προβλήματα να μην είναι εμπόδιο για την διεύρυνση. Ευχαριστώ κύριε Οσελ. Ο κύριος Μαυρονικόλα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο θέμα ενταξιακή πορεία, ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και Κυπριακών θα ήθελα να χαιρετήσω την καθαρή άποψη του κυρίου Επιτρόπου σε σχέση με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ένα, δύο σημεία τα οποία έχουν σχέση με τη δυνατότητα λύσης του κυπριακού προβλήματος και κατά πόσον η Επιτροπή σε ένα δεύτερο στάδιο θα πρέπει να επιληφθεί αυτών των θεμάτων. Είναι πρώτα η παρουσία του κατοχικού στρατού που νομίζω ότι και εσείς κύριε Επίτροπε είδατε το μέγεθος της παρουσίας αυτής σε ένα μικρό νησί και δεύτερο ο συνεχιζόμενος επικισμός από Τούρκους επίκους οι οποίοι μεταφέρονται στην ΕΦΟΣ στην Βόρεια Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε ένα ακόμα βήμα περισσότερο, ζητώντας από την Τουρκία, συμβάλλοντας ακριβώς για τις συνομιλίες, να αναλάβει ουσιαστική ρύθμιση, μείωση της κατοχικής παρουσίας και ελάττωσης των επίκοστων νησίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιγκολ για ένα λεπτό. Θα ήθελα να συγχαρώ και να πω ότι πραγματικά είμαι ικανοποιημένο με την έκθεση του Επιτρόπου και με τη γενική στάση της Κομισιόν. Καταδεικνύει ότι υπάρχει σταθερό ενδιαφέρον για διεύρυνση σαν μέσο πρόσθετης αξίας για τη, προς τη σταθερότητα της Ευρώπης. Θα περιοριστώ στα σχόλιά μου, στα καλά νέα για την Κροατία και το Μοντενέγκρο. Χαίρομαι που άκουσα αυτά τα καλά νέα. Έχουμε κακά νέα για την Αλβανία. Ίσως θα ήταν καλύτερα τα νέα από την Αλβανία αν διαχειριζόμασταν καλύτερα στο Ευρωκοινοβούλιο την πολιτική κρίση στην Αλβανία. Χωρίς να παίρνουμε το μέρος των αντιστοίχων κομμάτων εκεί, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να είμαστε διαμεσολαβητές για την επίλυση της πολιτικής κρίσης στην Αλβανία. Αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βάικολ. Ο κύριος Μπρίζατζιτς για ένα λεπτό. Η κυρία. Súhlasím s tým, čo pán Tanok povedal o Černej hore a prosím vás pre otvorenú a stručnú otázku. Čo je realistické za očakávať, kedy... Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω Ποιε μπορεί να είναι ε, ε, κάποιες ρεαλιστικές προσδοκίες. Πότε θα καλέσετε το Μοντενέγκρο για διαπραγματεύσεις. Ποια θα μπορούσε να είναι μια ρεαλιστική ημερομηνία. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κράιστοφλερ για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι οι υποψήφιε χώρε, οι δυνάμει υποψήφιε χώρε, όχι κράτη-μέλη, βρισκόμαστε σε μια ταύτιση υπολογιστή που έχει πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή του και θα λύσει όλα τα προβλήματα από μόνο του. Ενώ τα πράγματα είναι πολύ πολύπλοκα. Σας ρωτώ λοιπόν, αναφερθήκατε στο θέμα της δυνατότητας απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να υπάρχει. Πόσο ικανή θεωρείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα να δεχθεί άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτρελ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για τα σαφή λόγια που μας είπατε. Αυτό είναι ένα στοιχείο αξιοπιστία. Εγώ χαίρομαι για οποιαδήποτε πρόοδο. Εκεί που έχω πρόβλημα είναι με τις μεγάλες διαφορές ε, που υπάρχουν μεταξύ των χωρών τέος Ιουκοσλαβία. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει βέβαια το κράτος το ίδιο να καταπατά του, αλλά όπως είπαν και οι προλελήσαντες θα πρέπει να υπάρχουν πιο έντονες φιλοδοξίες, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε στις διαδικασίες που δημιουργούν καλύτερα ατμόσφαιρα, περισσότερη περιφερειακή συνεργασία και επίσης και ανατομικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα μπλοκαρίσματα που υπάρχουν που είναι ενοχλητικά και επικίνδυνα θα είναι πιο δύσκολο ίσως να καταρρύψουμε το τείχο στα Βαλκάνια από ότι το σιδερόν παραπέτασμα. Θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη φιλοδοξία και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε την διαδικασία αυτή. Είπαμε πάντα ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πέτρελε. Κύριε Σπότσκουτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω σύντομη ερώτηση. Εδώ είμαι κύριε Φούλα. Είπατε ότι μετά τις εκλογές θέλετε να πάτε στη Βοσνία για να παρακολουθήσετε τη διαργασία. Τι συγκεκριμένες ενέργειες έχετε κατά νου εκ μέρους της Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μεταρρυθμίσεις. Τουρκία. Α, επαναλάβετε την ερώτηση λέει ο κύριος Φούλα. Ναι, μιλάτε πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνω να σας καταλάβω. Ξαναρχίζω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Είπατε ότι μετά τις εκλογές θέλετε να πάτε στη Βοσνία για να παρακολουθήσετε εκ του σύνεγγυς τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικές για τη Βοσνία. Έχουμε λοιπόν την έκθεσή σας που το αναφέρει αυτό. Αλλά τι συγκεκριμένες ενέργειες προβλέπετε. Τουρκία τώρα, δεύτερη ερώτηση. Είμαστε σαν διαέξοδο με τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Είναι σημαντικές οι διαπραγματεύσεις και για τις δύο πλευρές. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν προβλέπει το ρόλο της, για να ποιο ρόλο θα αναλάβει για να ξεπεράσει αυτά τα διέξοδα. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Πενεραμπατού για ένα λεπτό. Α, συγγνώμη, έκανα λάθος. Κονέλησεν για ένα λεπτό, διορθώνει ο πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, ε, έκανα λάθος. Ο κύριος ε, η κυρία Κορνέλσεν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ως ε, εκπρόσωπος των Πρεσίνων για τη Βοσνία και ε, Ζεγοβίνη θα επικεντρωθώ σε αυτά τα θέματα. Όσον αφορά την Βοσνία, πολύ σωστά καλείται τους πολιτικού παράγοντε σε ενότητα. Ε, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το ίδιο πράγμα και να μιλήσει με μία φωνή προ τη Βοσνία. Κάποιοι θέλουν το α, κάποιοι θέλουν το αντίθετο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 κάποιοι κινούνται σε τοπικό επίπεδο χωρίς να ενημερώνουν το ομοσπονδιακό επίπεδο. Η αξιοπιστία λοιπόν ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θίγεται συνεχώς και πλήττεται από, την, ε, από τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ μας. Πρέπει να έχει μια ισχυρή φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεκινήσει πρωτοβουλίες για, την, ε, για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ε, όσον αφορά την Αλβανία, πραγματικά είναι χάλια τα πράγματα και συμφωνώ με τον κύριο Κάνι ε, και λέτε ότι προτείνεται να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ε, μόλις σταματήσουν να τρώγονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι σαφώς ε, στέλνετε την ευθύνη στη δική τους μεριά και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα που πρέπει να τους στείλουμε. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλισεν. Το λόγο έχει ε, ο κύριος Κόπα για ένα λεπτό. Η κυρία, με συγχωρείτε, Κόπα. Επίτροπο για τη σταθερή και συνεπή στάση του απέναντι στη διεύρυνση όλο αυτό το διάστημα. Θα μιλήσω ειδικά για το θέμα της Φύρομ και το θέμα του ονόματος που ετέθη από αρκετούς ε, συναδέλφους εδώ. Όλοι είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, αλλά για την επίλυση του ζητήματος πρέπει να γίνει σαφές ποιος επιθυμεί τη λύση και ποιος κολλησιεργεί. Όλο τον τελευταίο χρόνο η ελληνική κυβέρνηση έδειξε σε όλα τα επίπεδα ότι θέλει να κλείσει αυτό το ζήτημα, εγγενιάζοντας και τις επαφές σε επίπεδο πρωθυπουργών με εντατικές συζητήσεις με δική της πρωτοβουλία. Δυστυχώς δεν υπήρξε η ανταπόκριση που περιμέναμε. Ε, ο κύριος Γκρούευσκι δεν εμφανίστηκε στη συνάντηση της Νέας Υόρκης και αργότερα ζήτησε ο ίδιος και προκάλεσε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν διαπιστώνουμε όμως διάθεση για επίλυση και δυστυχώς δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι πραγματικά τον ενδιαφέρει να κλείσει αυτό το ζήτημα. Η ερώτηση μου είναι γιατί η Επιτροπή δεν καλεί συγκεκριμένα την κυβέρνηση των Σκοπίων να έρθει επικοδομητικά στο διάλογο αυτό. Από την ελληνική πλευρά νομίζω όλη η διάθεση είναι εμφανής. Ευχαριστώ κυρία Κόπα. Μπενερά Μπατού για ένα λεπτό. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της ένταξης της Τουρκίας είναι βασικό και για την Τουρκία και για την Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής. Η ολοκλήρωση μιας μουσουλμανικής χώρας βασικά στην Ευρώπη σημαίνει αναγνώριση των μουσουλμάνων πολιτών και του πλουραλισμού. Η ένταξη της Τουρκίας πρέπει να γίνει σε εύλογο χρόνο. Μετά από μια δεκαετία διαπραγματεύσεων πρέπει να βάλουμε μια προθεσμία λοιπόν. Όλα αυτά είναι σημαντικά Επίσης σημαντικό είναι η όρη αυτής της ένταξης. Αναφέρθηκε από τους συναδέλφους μου αυτό. Αναφέρομαι στην προστασία της πολι... πολιτισμικότητας της Τουρκίας. Σαν πράσινη είμαι για τα φράγματα, αλλά όταν χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού χωρίς να ρηπαίνουν. 19 υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην κουρδική περιοχή πρόκειται να οικοδομηθούν. Φράγμα στον Τίγρη, 45 χιλιόμετρα από την, τα σύνορα. Ε, έχουμε επιχειρήσεις πολλών κρασών που συμμετέχουν. κυρία Παπαδοπούλου ή ο κύριος Παπαδόπουλος. Με συγχωρείτε, δεν παρακολουθούμε πολύ εύκολα σήμερα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. In the progress report on Turkey, it is written that Turkey... Στην έκθεση πρώτου για την Κύπρο γράφει ότι η δέσμευση της Τουρκίας με συγκεκριμένου τρόπους για μια οριστική λύση στην Κύπρο έχει κρίσιμη σημασία. Κύριε Φούλε, συμφωνώ απόλυτα με την ε, δήλωση αυτή. Κατά τη γνώμη μου, η Κομισιόν δεν θα πρέπει να περιοριστεί να παρακολουθεί και να κάνει εκθέσεις μόνο για τη μη συμμόρφωση της ε, Τουρκίας με τις υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο να ζητηθεί από την Τουρκία να αποσύρει τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο και να σταματήσει τους παράνομους επικισμούς. Αυτό εννοείται όταν λέτε με συγκεκριμένους όρους. Σας παρακαλώ να το διευκρινίσετε. Μάλιστα, 29 ομιλητές πήραν το λόγο και πολλοί από αυτούς με περισσότερες από μία ερωτήσεις. Ξέρω ότι είναι πολύ πολύπλοκο το έργο του ε, Επιτρόπου ε, στην προσπάθεια του να απαντήσει. περιμένουμε απαντήσεις στο 100%. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί που σταματήσαμε στη συζήτησή μας. Δεν ήταν προς συμφέρον της Κομισιόν. Αναφέρομαι στην Τουρκία. Ε, δεν ήταν χρήσιμο για την Κομισιό να επαναλαμβάνει συνέχεια την επιμονή για την εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλου, του συμπληρωματικού πρωτοκόλου της συμφωνίας. Νομίζω ότι πέρυσι τα κράτη-μέλη το ε, κατέστησαν με μία αντίλωσή τους σαφή την κατάσταση σε σχέση με αυτό το ζήτημα της εφαρμογής του πρωτοκόλου. Πρόκειται για μια οδυνηρή διαδικασία που μας έφερε πράγματι σε μια κατάσταση όπου έχουμε μόνο τρία κεφάλαια προς διαπραγμάτευση και προς άνοιγμα και διαπραγμάτευση και για να μην χάσουμε την προθετική δύναμη, για να μην συγκρουστεί το, ε, το τρένο, θα έλεγα ότι είναι κατεπήγον για την Τουρκία να εφαρμόσει το ε, πρόσθετο πρωτόκολλο, το συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Κατεπήγον λοιπόν. Πράγματι, στις εφημερίδες διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι υπάρχουν μυστικές διαπραγματεύσεις. Δεν θα σχολιάσω τώρα αυτούς τους ισχυρισμούς του τύπου. Θα ήθελα να υποφεληθώ όμως από την ευκαιρία για να σας υπενθυμίσω τη δική μου θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι μυστικό ότι η Κομισιόν υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης στο Κυπριακό προς όφελος της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει, το είπα αυτό και προηγουμένως, να εφαρμόσει πλήρως το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Προσθέτω ακόμη ότι μαζί με τον συνάδελφο παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις σε σχέση με αυτά τα θέματα. Είμαι σε συνεχή επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς στους οποίους αναφερθήκατε. Uh, uh, uh, Κατόπιν πήγα στην Κύπρο και είδα και τους δύο ηγέτες εν δράση. Είδα να μιλούν προς τους Τούρκοκυπρίους, προς τους Ελληνοκυπρίους όταν άνοιξε το σημείο διάβαση και με εντυπωσίασε ο ενθουσιασμός ο ανοιχτό χαρακτήρας των πολιτών και από τις δύο πλευρές. Και βασιζόμενος σε συμπραγματικές συζητήσεις, εξασφαλίστηκε ότι τον συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για, τις, ε, για την τελική επίλυση και να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ότι αυτή η διαδικασία που προωθείται για τους δύο ηγέτες είναι εκείνη η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει αποτελέσματα κατά τον συντομότερο δυνατό τρόπο. Όχι, δεν είχα διαβουλεύσει εγώ με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά είχα ε, πολύ έντονη συζητήσει με τον κύριο Ντάουνερ, τον εκπρόσωπό του. Και ναι, είμαι σε επαφή μαζί τους και θα εξακολουθήσω να είμαι σε επαφή μαζί τους. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω ανοιχτό τρόπο διαπραγματεύσεων και όλα τα άλλα μέσα της ε, διπλωματίας για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την διαδικασία αυτή. Τώρα για την ίδια την Τουρκία. Δεν υπάρχουν πολλοί, ακόμα και στην διακεκριμένη αυτή επιτροπή τη δική σας, που είναι ικανοποιημένοι με τη βάση τον ε, διαπραγματεύσεων και το ρυθμό με τον οποίο προχωρούν. Δηλαδή ένα κεφάλαιο, ένα προεδρία. Αυτή τη στιγμή που είναι αρχές Νοεμβρίου δεν μπορώ καν να σας εγγυηθώ ότι θα ανοίξει ένα κεφάλαιο προς το τέλη του έτους. Χρειαζόμαστε μια νέα προθετική ορμή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε. Θα πρέπει να παραμείνουμε στη διαδικασία πλαίσιο, στην εντολή δηλαδή για την διαπραγμάτευση. Και έτσι θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Όχι όμως να μαχόμαστε για ένα κεφάλαιο ανά προεδρία και να αντιμετωπίσουμε το δίλημα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι ο καθαρός συσχετισμός με το συμπληρωματικό πρωτόκολλο είναι αυθερμοφανής. Και αυτό που είπε ο κ. Σαλαφράκα και άλλοι είναι επίση σωστό ότι όσο πιο μεγάλη πρόοδος υπάρχει στη σχέση μεταξύ Τουρκίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου θα επιταχύνει τη διαδικασία. Είναι σημαντικό Προσπαθώντας να βρούμε τη νέα αυτή προοδευτική ορμή στις διαπραγματεύσει να έχουμε σχέσεις με τους πιο δραστήριους παράγοντε της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Η είπατε εκπρόσωπος την πρόεδρος της Κομισιόν είναι σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας το θέμα αυτό, προσπαθώ να εξασφαλίσει ότι θα ωφεληθούμε από την ε, νέα αυτή αναγνώριση της σημασίας της ίδιας της Τουρκίας στην περιοχή εκεί. Να υπάρχει μια σχέση διαπραγματεύσεων με την Τουρκία όσον αφορά τα πιο κρίσιμα θέματα και δεν αναφέραμε μόνο στους άμεσους αλλά το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Και νομίζω ότι έχει κάθε συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να έχουμε και τις δύο διαστάσεις των σχέσεων αυτών με την Τουρκία. Αφενός δηλαδή η διαδικασία διευρυνση. που θα μας βοηθήσει να έχουμε λέγει σημαντικό και στην κατεύθυνση της διαδικασίας ε, μεταρρύθμισης στην ίδια την Τουρκία. Γιατί αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ωφεληθούμε από τις τουρκικές πολιτικές. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει και για την Τουρκία, η οποία ωφελείται από τις κοινωνικές αρχές και είμαι σίγουρος ότι και η ίδια η Τουρκία κατανοεί ότι όσο πιο πολλές σχέσεις έχουμε για το θέμα αυτό, τόσο πιο καλύτερα θα μπορεί να ανεκατοπτρίσει στην εξωτερική της πολιτική τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η διαδικασία διάβρυνσης. Uh, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, της Μακεδονίας. Δεν έχω χάσει τον ενθουσιασμό μου στη σχέση με αυτή τη χώρα το, πλαίσιο και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαπραγματευτών και των δύο πρωθυπουργών μπορεί να επιφέρουν τελικά λύση και μεταβολή όσον αφορά την ονομασία. Ειλικρινά, δεν θέλω να εμπλακώ στη συζήτηση για το ποιος θα πιεστεί παραπάνω και ποιος λιγότερο. Νομίζω ότι και οι δύο πρωθυπουργοί αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Παπανδρέου, αντιλαμβάνεται πόσο αυτό το θέμα είναι μέρος του οράματος των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη. Και ο κύριος Γκρουεύσκη επίσης καταλαβαίνει σαφέστατα ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β για τη Φύρομ. Είμαι... Έχω τακτικές επαφές με τα μέρη. Αν αισθανθώ, πιστέψτε με, ότι υπάρχει λογικός χώρος για κάποιον άλλον παρεμβαίνοντα, δεν θα διστάσω μαζί με τον πρόεδρο Μπαρόσο. Δεν θα διστάσω να προσφέρω συγκεκριμένη βοήθεια. Συνεπώς η βοήθεια είναι διαθέσιμη και χορηγείται με πολλές μορφές. Αλλά όσο χρόνο αυτή η διαδικασία ε, είναι στα χέρια των Πρωθυπουργών. Παραμένω αισιόδοξο. ότι κάπου στο εγγύς μέλλον θα εξευρεθεί λύση. Και τώρα, για να οργανωθώ λίγο, μου λείπει σελίδα 4 από τις μειώσεις μου, τη βρήκα. Ωραία. Όσον αφορά την ημερομηνία για την Κροατία, για την κατάληξη της, των διαπραγματεύσεων ένταξης, δεν μπορώ σοβαρά να επικεντρωθώ στην αξιοπιστία και ταυτόχρονα για τρίτη συνεχή χρονιά να επαναλαμβάνω ότι του χρόνου θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Ξανά το ίδιο πράγμα από χρόνο σε χρόνο. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Όχι. Αντίθετα, η Κροατία έχει πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο. Αλλά το τελευταίο άλμα καμιά φορά είναι το πιο δύσκολο. Ξέρετε, τα δύσκολα σημεία του κεφαλαίου 23 που αφορά το ιστορικό της διαδρομής και υπάρχουν ορισμένα benchmarks τα οποία αντιμετωπίζει η Κροατία. Είμαι ε, σίγουρος ότι οι αρχές της Κροατίας αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του κεφαλαίου 23. Καταλαβαίνουν επίσης και την προσέγγιση της Κομισιόν. Ξέρουν από τον συνεχή μας διάλογο ότι το Μάρτιο του χρόνου θα αξιολογήσουμε την εφαρμογή αυτών των benchmarks. Και τότε θα είμαστε σαφέστεροι ως προς την χρονική στιγμή. Αλλά ως προς τη θεωρητική ερώτηση, αν είναι ρεαλιστικό κάτω από τους συγκεκριμένους όρους ε, να, καταλήξει να, καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις κάτω από Ουγγρική Προεδρία. Ναι, είναι εφικτό. Θεωρητική ερώτηση, θεωρητική απάντηση. Θα μπορούσε βεβαίως να είναι και η Πολωνική Προεδρία που θα διαδεχθεί την Ουγγρική. Αλλά υπάρχουν όροι. Συνεπώς, η ημερομηνία είναι στα χέρια των Κροατών, των αρχών της Κροατίας και των πολιτών. Μοντενέγκρο τώρα. Πότε θα μπορέσει να έχει ημερομηνία για διαπραγματεύσει ένταξη στο Μοντενέγκρο. Και σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω ότι είμαστε στα χέρια του Μοντενέγκρο, του Μαυροβουνίου και έτσι απαντώ και σε μια από τις ερωτήσεις. Δεν επινοήσαμε εμείς ή, ή, δεν γυρίσαμε τη μακεδονική υπόθεση σε θέση, ε, ε, σε τοποθέτηση ευρωπαϊκή, δηλαδή ε, θα έχετε καθεστώς υποψηφίου αλλά δεν θα έχετε διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν 7-8 χώρες που αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση. Δηλαδή δεν αναφέρεται αυτό μόνο στη Φύρο. Στη Μακεδονία. Η ημερομηνία των διαπραγματεύσεων είναι στα χέρια του Μαυροβουνίου. Σε μεγάλο βαθμό. Τους βοηθήσαμε. δίνοντας 7 προτεραιότητες κλειδιά προς εφαρμογή. Μόλις λοιπόν πραγματοποιήσουν την υλοποίησή τους και συνεχίσουν την θετική τους τροχιά και σε άλλα θέματα, υλοποιήσουν τη σταθεροποίηση, την συμφωνία προσχώρησης κτλ. Τότε η Κομισιόν θα μπορέσει να γίνει πιο συγκεκριμένη. Αλλά το ίδιο ισχύει και για την Αλβανία άλλωστε. Το γεγονό ότι δεν είμαι σε θέση ή έτοιμος μάλλον σε αυτή τη φάση να προτίσω στους συναδέλφους της Κομισιόν και σε εσά το καθεστώς υποψηφίου για την Αλβανία, αυτό δεν σημαίνει ότι η Αλβανία δεν μπορεί να βρεθεί στην ίδια κατάσταση όπως αυτή που μόλις περιέγραψα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι στα χέρια των χωρών τελικά. Ελέγχθη ότι ίσως δεν έχουμε τα πολύ αποτελεσματικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε τη διεύρυνση. Θα, θα είχα αντίρρηση γι' αυτό. Θα έλεγα ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε την διεύρυνση και να προσθέσουμε και ένα πολιτικό στοιχείο, μια πολιτική κατεύθυνση. Δηλαδή, συμφωνώ με όσους λένε εδώ ότι η διεύρυνση δεν πρέπει να είναι απλώς μια τεχνική άσκηση. Και ότι πράγματι είναι μια πολιτική διαργασία πολιτικά σημαίνουσα διαδικασία. Συνεπώς πρέπει να καθοδηγείται και πολιτικά. Και η διάδραση με το Ευρωκοινοβούλιο, η οποία μου είναι ευπρόσδεκτη, δίνει στην Κομισιό και σε μένα και ενδεχομένω και στο Συμβουλίο τη δυνατότητα να καθοδηγήσουμε πολιτικά αυτή τη διεργασία. Πόση ικανότητα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά, ε, πόση χωρητικότητα θα λέγαμε, ε, πόσο μπορεί να απορροφήσει νέα κράτη-μέλη. Θα είμαι απολύτως σαφής. Δεν έχω κατά κανέναν τρόπο πρόθεση να αναφέρω ότι υπάρχουν κάποια θεσμικά ε, σημεία συμφόρησης ακόμα. Τα έχουμε φροντίσει αυτά τα θέματα και έχουμε ανοίξει την πόρτα προς τις ε, υποψήφιες χώρες και στις χώρες που ευελπιστούν να γίνουν υποψήφιες για να περάσουν από αυτή την πόρτα. Τώρα, όμως, το κατά πόσον ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100% έτοιμη να υποδεχτεί την κάθε υποψήφια χώρα, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποψήφια χώρα. Εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις. Θα εξαρτηθεί τι θα γίνει κατά το χρόνο πριν από τη λήψη της απόφασης. Πώς θα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο που θα έχει η ένταξη της κάθε συγκεκριμένης υποψήφιας χώρας ε, και ποιος είναι ο αντίκτυπος πάνω στις συγκεκριμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ε, ε, υπάρξει συνομιλία βεβαίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Για την Βοσνία Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό που καταφέραμε ε, αμέσως μετά τις εκλογές να στείλουμε αυτό το μήνυμα ε, λέγοντας ότι όποια και η συμμαχία και το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να είναι ευρωκεντρικό το πρώτο και δεύτερον ότι θα πρέπει να ε, γίνει σαφές ποιες είναι οι προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έρθει η χρονική στιγμή ε, μετά το σχηματισμό της ε, κυβερνητική ε, συμμαχία. ελπίζω, λέω, ότι θα έρθει η στιγμή να σεβαστούν τι δεσμεύσει του. Και εγώ μαζί με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ε, από το γραφείο ε, της ΕΠΑ της ε, σε ενισχυμένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πορεία προς την κατεύθυνση ενός λειτουργικού κράτους το οποίο στη συνέχεια θα μας δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε σημαντικά βήματα στη διαδικασία διεύρυνσης. Στα συμπεράσματα και στις συστάσεις θα δείτε ότι υπάρχει μια σημαντική αναφορά στην Ευρώπη ε, του 2020. Και πάλι αυτό είναι κάτι που είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρώπη 2020 είναι το πρώτο τέτοιο στρατηγικό έγγραφο της Κομισιόν που έχει μια εξωτερική διάσταση. Και στα συμπεράσματά μας και στις συστάσεις μας καλούμε τις υποψήφιες χώρες και τις ε, που ευελπιστούν ε, να ε, ε, προβληματιστούν σχετικά με τους στόχους του ε, γράφου μας αυτού και της ενσωμάτωσής τους στα δικά, τους προγράμματα. Και ελπίζουμε ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία, η στρατηγική δηλαδή του 2020. Για την Ισλανδία... Νομίζω ότι υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Υπάρχουν, ε, υπάρχει το θέμα των ε, πόρων uh, του προενταξιακού μέσου, καταρχάς, ε, που θα πρέπει να βελτιώσει τις διοικητικές ικανότητες και θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων εν ώψη της ε, ένταξης και φυσικά ε, το μέσο αυτό θα ε, βελτιώσει την ικανότητα του κράτους στο μέλλον να διαχειριστεί τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτός είναι ο ρόλος του προενταξιακού μέσου. Ταυτόχρονα, όπως βλέπουμε την σταδιακή αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεται η, Ευρωπαϊκή, η κοινή γνώμη την Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούμε με συγκεκριμένες πράξεις για να, κάτι, να απαλείψουμε ε, κάποιες παρανοήσεις όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, γι' αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί οι πόροι για την ε, πολιτική επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι οι διερμηνείς θα περιμένουν να σταματήσω όπου να είναι, γι' αυτό θα σταματήσω τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι αυτή ε, η συνάντηση σήμερα είναι το τέλος των συνομιλιών μας για αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν με αυτή τη μορφή ή ε, στο πλαίσιο ε, συνομιλιών κατά την Ολομέλεια του Στρασβούργου. Δεν ξέρω με ποια μορφή θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Θα το αποφασίσετε εσείς αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εμείς ε, αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι η συζήτησή μας θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση ε, με την οποία ξεκίνησε. Εκτιμούμε όλη αυτή την συνεργασία. 18 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, με συγχωρείτε στις Βρυξέλλες, είναι η επόμενη ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πέρα στις συνεδρίαση